Okay, we, um, we continue. We actually start with our, with our seminar for today. Ξεκινάμε το σεμινάριο μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω εδώ στην Ευρώπη της Ασυλία Βέξτρομ, βουλευτή της ομάδας ALDE και από τη Σουηδία. Η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Έχετε τον λόγο για να μας μιλήσετε για την εκθεσή σας. Το βασικό ερώτημα που θα έκανα εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος θα ήταν για ποιο λόγο είναι σημαντικό το θέμα αυτό και για ποιο λόγο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Οπότε σας δίνω το λόγο να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να νιώσετε ότι η εκδήλωσή μας ε, απαντάει στις ε, ανησυχίες των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι η Σεσίλια Βίκστρομ, είμαι φιλελεύθερη από τη Σουηδία και είμαι η για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός του Δουβλίνου είναι ένα από τα νομοθετικά ε, μια από τις νομοθετικές ε, πράξει που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Οι σκιώδει εισηγητές μου, δηλαδή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν ε, τις άλλες πολιτικές ομάδες στην διαπραγματευτική μου ομάδα, είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία και νομίζω ότι κάποιοι από, εδώ, κάποιοι από αυτούς είναι παρόντε, θα έπρεπε να είναι. Έχουμε ασχοληθεί με την πρόταση αυτή εδώ και αρκετό καιρό και υπέβαλα σχέδιο έκθεσης με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν οι συνάδελφοι υπέβαλαν πάνω από χίλιες τροπολογίες. Νέες προτάσεις δηλαδή τροποποίησης του κειμένου μου να γίνει πιο σαφές. Και τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις πάνω σε κάθε άρθρο μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και Αφού το κάνουμε αυτό, θα έχουμε ολοκληρώσει λίγο πολύ την αποστολή μας, διότι έτσι θα έχει διαμορφωθεί η θέση του Κοινοβουλίου και θα είμαστε πια έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δηλαδή με το Συμβούλιο Υπουργών, τους εκπροσώπους των κρατών μελών. Και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο το όλο θέμα, διότι όπως γνωρίζετε οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συναντούν δυσκολίες στον τομέα αυτών του ασύλου, δηλαδή και της μετανάστευση όσον αφορά την ε, εξέβρεση κοινή θέση. Ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ εύκολο να βρεθεί κοινή θέση. Στο Κοινοβούλιο όμως είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες μας και να καταλήξουμε σε κοινή θέση. αφού το Συμβούλιο καταλήξει σε κοινή θέση, σε μια ενιαία θέση, πολύ ευχαριστώ, ε, θα συμμετάσχω σε τριμερή διάλογο και θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Θα καταλήξουμε σε συμφωνία στο θέμα αυτό. Εφόσον το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο καταφέρουν να συμφωνήσουν πάνω σε ένα κείμενο. Εδώ στο Κοινοβούλιο απαιτείται πλειοψηφία, στο Συμβούλιο απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται όμως ομόφωνη απόφαση, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να υιοθετηθεί η θέση τους. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, στις οποίες θα είμαι η θα ξεκινήσουν μετά το ε, καλοκαίρι, αφού επιστρέψουμε από τις διακοπές. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Το Κοινοβούλιο δεν θα δεχτεί τρελές ιδέες από τα κράτη-μέλη. και δεν θα δεχτεί πρόταση που να μην αλλάζει την πραγματική κατάσταση, διότι όπως γνωρίζετε το 2015 κατέρευσε το σύστημα. Είδαμε ανθρώπους να καταφθάνουν στην Ευρώπη από διάφορες οδούς. Είδαμε εικόνες στην τηλεόραση, τις οποίες δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Νομίζω ότι ε, είναι μια θέση που ε, συμμερίζεστε κι εσείς να επικεντρωθώ αυτή τη στιγμή σε κάποια στοιχεία της πρότασης. Όλοι συμφωνούμε ότι το ισχύον σύστημα δεν λειτουργεί. Έχει καταρρεύσει ακόμα και τα κράτη-μέλη, ακόμα και το Συμβούλιο συμφωνεί σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου απέτυχε το τεστ της πραγματικότητας το 2015. Και να σας πω την αλήθεια, ούτε και πριν λειτουργούσε Πρέπει λοιπόν να πούμε δυνατά ότι πρόκειται για αποτυχία. Και αν συνεχίσουμε να επιμένουμε τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής, η Ελλάδα και η Ιταλία για παράδειγμα, να φέρουν όλο το βάρος ε, και τον κίνδυνο, το σύστημα αυτό δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κανένας ε, των άσυλο να μην καταχωρείται, όπως είδαμε το 2015, και οι άνθρωποι να μετακινηθούν μόνοι του προς τον προορισμό που θέλουν. Και πριν την κρίση, ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν λειτουργούσε σωστά. Οι εργασίες πάνω στον κανονισμό αυτό ε, ξεκίνησαν το 1999 και είναι πρόταση που δεν ε, ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκες του σήμερα. Ακόμα και πριν το 2015, το 3 ή 4% μόλις των ετούντων άσυλο μεταφέρονταν σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Το σύστημα λοιπόν ε, είναι πια νεκρό. Ήταν στην εντατική μάλλον τα τελευταία χρόνια, τώρα πια είναι νεκρό όμως. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί, ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις βασικές αρχές της Σύμβασης της Γενέβης ε, και του ασύλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε ζητάει ασύλο θα, ε, ε, το, θα έχει δικαίωμα να το λάβει εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Επίσης, όσοι δεν πληρούν τις υποθέσει θα πρέπει να επιστρέφονται. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, στον κανονισμό του Δουβλίνου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κάποια βασικά στοιχεία. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να φροντίσουμε κάθε κράτος μέλος να φέρει δίκαιο μερίδιο της ευθύνης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από ε, πέντε κράτη-μέλη από τα 28 να φέρουν όλο το βάρος. Η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι μόνιμο στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής ε, του κανονισμού του Δουβλίνου. Συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και είναι ένα θέμα το οποίο έχω τονίσει ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε οι οικογένειες να παραμένουν ενωμένες και να λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις ε, του ετούντα με κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ε, εάν υπάρχουν. Και άνθρωποι που έχουν συνταξιδέψει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορούν επίσης να ε, παραμείνουν μαζί. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε ο κάθε ετών να λαμβάνει σωστές πληροφορίες και να υπάρχουν εγγυήσει ιδιαίτερα για τα παιδιά και, τα, και τους ασυνόδευτούς ανήλικους. Έτσι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα από τη μία από την πλευρά των ετούντων και από την άλλη από την πλευρά των κρατών μελών. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης οι ετούντες θα πρέπει να παραμένουν στο κράτος μέλος το οποίο έχει αποφασιστεί ότι είναι αρμόδιο για την ε, απόφαση περί ασύλου. Σήμερα υπάρχουν πολλά παραθυράκια στο σύστημα, επιτρέπουν στους ετούντες ε, να μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος και έτσι να υπάρχει μεταφορά της ευθύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό όμως θα πρέπει να σταματήσει, διότι αλλιώς θα συνεχίσουν ε, ελάχιστα κράτη-μέλη να κάνουν όλη τη δουλειά και τα υπόλοιπα να μην κάνουν τίποτα. Βλέπουμε δευτερογενεί κινήσεις σήμερα, διότι είναι αδύνατον ε, να εφαρμόσουμε ένα σύστημα όπου οι ετούντε να παραμένουν εκεί που πρέπει, διότι το σύστημα ενθαρρύνει τους ετούντε να μετακινηθούν σε άλλο μέρος ε, ή να μετακινούνται κάτω από το ραντάρ, ώστε να μην ε, τους εντοπίζουν οι αρχές απόφαση στο Συμβούλιο απαιτεί ειδική πλειοψηφία και αφού ληφθεί κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να σεβαστεί την απόφαση αυτή. Έτσι νομοθετούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να το κάνουν αυτό ακόμα και αν έχουν ε, καταψηφίσει την πρόταση. Δεν είναι μπουφές ε, το η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μπορεί κανείς να επιλέγει ποια στοιχεία θέλει να πάρει. Προτείνω όμως ένα σύστημα όπου εάν κάποιο κράτος μέλος δεν θέλει να εφαρμόσει το σύστημα να μπορούν να παρακρατηθούν κάποιοι πόροι από τα διαστροτικά ταμεία για παράδειγμα. Αυτό δεν θα γίνει εφόσον τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόσουν το σύστημα και σεβαστούν ε, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πάνω στην πρόταση αυτή. Μα περιμένει όμως μακρύ ταξίδι. Είμαι πεπισμένη ότι στο Κοινοβούλιο θα καταλήξουμε σε ευρία πλειοψηφία πάνω σε μια ρεαλιστική και φιλόδοξη πρόταση που θα αλλάξει την κατάσταση. Θα έχουμε ανοιχτέ διαπραγματεύσει. Ε, θα ε, είμαι εγώ επικεφαλής στις διαπραγματεύσει με τις κυβερνήσει των κρατών μελών. Όμω, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα σύστημα το οποίο θεωρούμε ότι θα αποτύχει. Εάν δεν αλλάξει την κατάσταση, το νέο σύστημα δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε και να εγχωρίσουμε μόνο και μόνο για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα πρέπει να φροντίσουμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα να αλλάζει την σημερινή κατάσταση και να καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν επί ίσης και να αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο της ευθύνης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομοθετήσει την αλληλεγγύη, μπορεί όμως να νομοθετήσει ώστε στην πραγματικότητα να οικοδομηθεί ε, ε, αλληλεγγύη και σε αυτήν τη θέση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι, δεσμευόμαστε να καταλήξουμε σε μία λύση που θα οδηγήσει σε αλληλεγγύη. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Mrs. That was very lucid and clear. Ευχαριστώ κυρία Βίκτρομ, Ήταν σαφέστατη και διαυγής στην παρουσίαση αυτή. Ε, θα ακούσουμε τώρα δύο-τρεις ερωτήσεις και στη συνέχεια ε, θα έχουμε μια πρώτη απάντηση και μετά και άλλες ερωτήσεις. Υπάρχει διερμηνία, σας θυμίζω, οπότε μπορείτε να θέσετε ερωτήματα είτε στα αγγλικά, είτε στα γαλλικά, είτε στα γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά και σουηδικά, καθώς και βουλγάρικα. Ε, καλό είναι επίσης να μας ε, συστήνεστε πριν θέσετε το ερώτημά σας και επίσης σας παρακαλώ να μιλάτε αργά. Λοιπόν, κάποιος ζητάει το λόγο εκεί πίσω. Παρακαλώ. Ναι, Είμαι από την Εστονία. Το όνομα μου είναι Κόριν Κρέσσαλ, Εργάζομαι σε μια εφημερίδα τοπική για τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Ε, η χώρα μου έχει υποδεχθεί μια σειρά από πρόσφυγες. Όμως όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον οι μισοί έχουν ήδη φύγει. Ε, στην Λετωνία μπορεί να είναι και περισσότεροι αυτοί που έχουν φύγει. Είμαστε σε ένα καθεστώ δημοκρατία, ανοιχτών συνόρων. Πώ μπορούμε να του αποτρέψουμε από το να το κάνουν αυτό. Thank you very much. else. Ευχαριστώ. Άλλε ερωτήσει. Ε, όχι. Ναι, παρακαλώ. Το όνομά μου είναι Μιχαλ Κόκολ από την Πολωνία. Χθε η τσεχική κυβέρνηση αποφάσισε να μην ε, υποδεχθεί κανέναν πρόσφυγα με βάση την απόφαση των τεσσάρων χωρών πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ε, ε, ε, συμφωνία στο Κοινοβούλιο, είπαμε, Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία έχουν ε, πει ότι δεν θα δεχτούν κανέναν επιπλέον Πρόσφατα και χθε μάλιστα η Τσεχή κυβέρνηση με την απόφασή τη. Ε, ωραία, απαντήστε σε αυτά τα ερωτήματα ήδη. Λοιπόν, ακούστε για την κατάσταση σχετικά με τι δευτερογενεί μετακινήσει. Είμαι σε διάλογο και με τον Υπουργό σας τον, από την Εστονία. Θα αναλάβετε μάλιστα την Προεδρία μετά τη Μάλτα, από τον Ιούλιο και μετά. Η Εστονία λοιπόν είναι αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και ε, αναμένω μια ε, θαραλέα Προεδρία, ε, διότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ο Υπουργός με τον οποίο μίλησα έχει την θέληση που έχω και εγώ για να προχωρήσουμε από ό,τι φαίνεται σε ό,τι αφορά τώρα την αποφυγή των δευτερογενών μετακινήσεων. Ακούστε, εάν δεν κάνουμε τίποτα, εάν δηλαδή το αφήσουμε αυτό να συμβαίνει, δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο όπου ουσιαστικά μια χούφτα χωρών είναι αυτή που υπομίζεται όλο το βάρος. Οι περισσότεροι δεν θα κάνουν τίποτα και θα παρακολουθούν απλώς τα Αυτό που λοιπόν πρέπει να κάνουμε είναι να, να εναρμονίσουμε την νομοθεσία. Δηλαδή, οι οδηγίες να ε, μετατραπούν σε κανονισμούς. Το επίπεδο προστασίας είναι υψηλό. Οι συνθήκες υποδοχής, οι προδιαγραφές είναι αρκετά καλές παντού. Αυτό, πρέπει να είναι ο στόχος μάλλον πρέπει να ε, δημιουργήσουμε αυτές τις, ε, αυτή τη διασπορά ε, παντού. Να το αφήσουμε να συμβεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου. Στη Σουηδία τη χώρα μου πριν από 130 χρόνια περίπου 25% του πληθυσμού τότε έφυγε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έμειναν στο Ellis Island και στη Νέα Υόρκη, πήγαν και στη Μινεάπολη, πήγαν μέχρι το κέντρο της Υπήρου και εκεί έφτασαν τα χωριά τους. Έφτιαξαν τα χωριά τους ε, από τις ίδιες γειτονιές, από τις ίδιες οικογένειες, από τα ίδια σχολεία, συμμαθητές. Υπήρχε μια διασπορά λοιπόν Σουηδών. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχουν, υπάρχει διασπορά Σύριων στην Γερμανία, στην Αυστρία, στη Σουηδία και αλλού. Αλλά όχι στην Κροατία και ίσως όχι και τόσο στη Λιθουανία Θα πρέπει λοιπόν να το εξασφαλίσουμε αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους, οποίους να γνωρίζουν εκεί. Χρειαζόμαστε πάντως κυρίως ένα αρμονισμένο σύστημα που το επίπεδο προστασίας είναι επαρκές, είναι αποδεκτό. Αυτό είναι που θα μας οδηγήσει στο να αποφύγουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Δηλαδή λέτε ότι το σύστημα, δεν, το σύστημα μας δεν είναι αρκετά καλό αυτή τη στιγμή. Το σύστημα δεν είναι αρκετά καλό πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Είναι κακό. Να σα πω την αλήθεια, οι χώρες οι οποίες έχουν δεχτεί περισσότερου μετανάστες το 2015, η Σουηδία και η Γερμανία δηλαδή, ε, εκεί ίσως να είναι και χειρότερη κατάσταση από ότι οπουδήποτε αλλού. Διότι η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Πρέπει να περιμένουν πολύ καιρό, διότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Δεν μπορούμε λοιπόν να δακτυλοδείχνουμε τον ένα και τον άλλον, να λέμε ότι ο ένα είναι καλό και άλλο κακό. Μαζί, μαζί πρέπει να κινηθούμε. Αυτό είναι το κλειδί. Και θα πρέπει να υπομισθούμε τι ευθύνε μα όλοι μαζί. Να απαντήσω τώρα στον Πολωνό φίλο για την τσεχική κυβέρνηση και του πρόσφυγε ε, και αυτό που είπατε, γιατί είπατε, αναφέρατε, στι χώρε του Βίζεγκραντ, οι οποίε από κοινού είπαν ότι εμεί δεν θέλουμε πρόσφυγε στο έδαφο μα. Ευτυχώς, οι χώρες του Βίζεγκραντ δεν μπορούν να μπλοκάρουν μια απόφαση. Το Συμβούλιο δεν χρειάζεται να πάρει απόφαση ομόφωνα. Μια ενισχυμένη πλειοψηφία αρκεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η επόμενη Προεδρία θα φανεί θαραλέα. Ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις. Εσείς πίσω. Ποιος άλλος. Ο κύριος εκεί και η κυρία εδώ. Μπρόχα, German News Agency. Θα ήθελα να πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Πριν μερικέ εβδομάδε είπατε ότι είστε αισιόδοξοι ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτου με ψηφοφορία στην Επιτροπή. Πότε πιστεύετε ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει την ψηφοφορία στην Επιτροπή Λίμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος εδώ. Ε, Σαλβατόρε Ντικάστρια, ε, πρακτορείο τύπου, Ιταλικό, Σαλβατόρε Λικάστρα, την Ατζεντσία της Στάμπα, Ιταλ Press, ε, από τη Σικελία. θωριακή περιοχή που βρίσκεται μέσω μιας θάλασσας που δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια είναι μια θάλασσα δυστυχίας. Αυτή η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου πώς μπορεί να περιορίσει την ανθρωπιστική τραγωδία και πώς θα λάβουμε υπόψη την βούληση των των ασυλών να επανενωθούν με τους συγγενείς και φίλους τους. Υπάρχει βούληση για να θέσουμε τέλος σε ένα σύστημα top-down το οποίο δεν λαμβάνει σε καμία περίπτωση υπόψη τις δικές τους ανάγκες αλλά βασίζεται σε απλά μαθηματικούς υπολογισμούς. Και τι θα γίνει με το τιμωρητικό του σοφρονιστικό σύστημα προς χώρες που αρνούνται να δεχθούν ετούντες άσυλο ανεξαρτήτως υπολογισμών και αριθμών. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ εσείς. Εστέρ, από την ε, Εφημερίδα Ραθιών στην Ισπανία. Θα ήθελα να μου πείτε το σύστημα ποσοστώσεων θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά το καλοκαίρι διότι κάποιες χώρες ε, τα πάνε καλά, άλλες όχι. Θα υπάρξουν πρόστιμα για αυτές τις χώρες διότι κάποιες είναι πιο υπέρ των προσφύγων και άλλες λιγότερο. Αυτό, ευχαριστώ. floor is Έχετε το λόγο. Κύριε Βίξτρο, με ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαμε να χτυπηθούμε στη δουλειά και να σας δώσουμε ένα κείμενο. Αλλά δεν έχει νόημα να βιαζόμαστε. Όπως ξέρουμε, το Συμβούλιο επίσης ε, χρονοτριβεί. Ρεαλιστικά, το χρονοδιάγραμμα θα, θα μπορούσε να είναι τέτοιο που ίσως και πριν τις θερινές διακοπές να έχουμε ήδη μια θέση του Κοινοβουλίου. Σαφή. Ενώπιον της Επιτροπής Λίμπε. είτε ακριβώς πριν είτε ακριβώς μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και όπως καταλαβαίνετε και είναι αυτονόητο, δεν είναι κάτι εύκολο, καθόλου μάλιστα, αλλά ρεαλιστικό, απόλυτα. Αλλά χρειάζεται συνεργασία. Όταν οι ομόλογοι μου λοιπόν στο άλλο θεσμικό όργανο δεν κινούνται ιδιαίτερως, Ξέρετε, μου λένε υπάρχουν πολλέ ε, ομάδε εργασία, πολλέ προτάσει νέων κειμένων για την ελληνική και ένα σωρό ε, χαζομάρε, ε, κείμενα τα οποία ανήκουν στον καλωθό των αχρήστων και όταν είναι έτσι πρέπει να ξεκινάει κανεί τα πράγματα πάλι από την αρχή Οπότε ελπίζουμε τώρα στην επόμενη Προεδρία να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα δείξουν θάρρο και θα αφιερώσουν και θα επενδύσουν κάποιε ώρε εργασία αποτελεσματικέ για να καταλήξουμε σε κάτι που θα λειτουργήσει την πραγματικότητα, που θα αλλάξει την πραγματικότητα. Προ το Σικελόφιλο έχω πάει στου προσφυγικού καταβλισμού στη Σικελία και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στη Σικελία, στη Λαπεντούζα Φυσικά οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν το δικαίωμα επανένωση με τους συγγενεί τους. Αυτό είναι αυτονόητο. Πριν από οποιοδήποτε δουβλίνο, στην πρότασή μου θα πρέπει να έχει προτεραιότητα η οικογενειακή επανένωση. Επίσης θέλω να δώσουμε τη δυνατότητα οι διακριτικές ρήτρε να δραστηριοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν. Είναι ένα καλό εργαλείο ε, που δείχνει τις συνάφειες ενός ανθρώπου με μια χώρα, αν έχει κάποιες γλωσσικές γνώσεις, κάποια έχει ενδεχομένως να ακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή έχει εργαστεί σε μια περιοχή, σε μια χώρα, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα όλα αυτά τα επιχειρήματα να τα χρησιμοποιήσει για να ζητήσει να πάει σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Να κάνει την αξιολόγηση τη αίτηση ασύλου η χώρα αυτή. Και το κίνητρο για μια τέτοια χώρα θα ήταν σε αυτή την περίπτωση μεγάλο, διότι ανάλογα με το μηχανισμό ε, κατανομής θα μπορούσαν, θα έπρεπε ούτω ή άλλω να πάρουν κάποιου γιατί να μην πάρουν αυτού οι οποίοι ρητά έχουν ζητήσει τη συγκεκριμένη χώρα. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο ε, ανάδειξη τη συνάφεια ε, ενό ατόμου με κάποια χώρα. Τώρα, όσον αφορά τι ποσοστώσει, αν θα υπάρξουν πρόστιμα, αν θα υπάρξουν άλλε συνέπειε. Κοιτάξτε, είναι αδιαμφισβήτητο ότι όταν δεν συμμορφώνεται κάποιος με το σύμφωνο χρηματοοικονομικής σταθερότητας, αυτό συνεπάγεται κάποιες οικονομικές συνέπειες. Αλλά σε αυτό το τομέα πολιτικής, τα κράτη-μέλη φαίνεται να θεωρούν ότι πρόκειται για ένα μπουφέ, όπου επιλέγουν να φάνε ό,τι θέλουν. Εφόσον θα υπάρχει λοιπόν νομοθεσία μέσω μια μεικτή διαδικασία, ε, μια κοινή διαδικασία με του συνομοθέτε και εφόσον έχουμε καταλήξει ένα κείμενο κοινώ αποδεκτό, τότε θα πρέπει να συμμορφώνονται άπαντε. Αυτό ισχύει για την ενέργεια, για την περιβαλλοντική νομοθεσία, ε, για τα χημικά, για οτιδήποτε. Φυσικά πρέπει να τηρεί κάποιου κανόνε, όλοι. Και όποιο δεν του τηρεί θα πρέπει να υφίσταται συνέπειε. Ωραία λοιπόν, ο κύριος εδώ, ο κύριος εκεί και η κυρία πιο πίσω. Ευχαριστώ. Uh, uh, from Slovakia, from... Γεια σας, από τη Σλοβακία. Η κυβέρνησή μας αρνήθηκε να δεχτεί ποσοστώσεις προσφύγων. Πώς βλέπετε την πολιτική βούληση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι το σύστημα απέτυχε και ότι πρέπει να τροποποιηθεί το σύστημα. Υπάρχει η υποστήριξη από την πλειοψηφία κατά των τεσσάρων κακών χωρών εντός εισαγωγικών. Ε, η Δανία, οι κάτω χώρες πιστεύετε ότι θα συμφωνήσουν και πιστεύετε ότι εντός του έτους θα υπάρξει σχετική απόφαση. Γεια σας. Ε, είπατε ότι οι συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες θα πρέπει να είναι καλές σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν ιδίου είδους υποστήριξη σε όλα τα κράτη. Επίσης είπατε ότι οι τέσσερις χώρες του Βίζεκράτ δεν ε, είναι αρκετές για να μπλοκάρουν την απόφαση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει λέγει στο θέμα αυτό. Ε, οι, κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ από την Ισλανδία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την ένταξη διότι οι δυτικέ χώρες ε, φοβούνται όλο και περισσότερο τους ε, πρόσφυγες. Ε, το είδαμε στο Λονδίνο, το Σαββατοκύριακο, το έχουμε δει και στο Παρίσι. Τι μπορεί να γίνει για να προωθηθεί η ένταξη των ανθρώπων αυτών και αυτοί οι ίδιοι που καταφτάνουν τι μπορούν να κάνουν από τη δική του πλευρά, διότι η ένταξη στην κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, ε, φαίνεται οι χώρες του Βίζεγκραντ να ε, ε, είναι οι πιο ξύπνιες μέσα στην αίθουσα αυτή. Στον κύριο από τη Σλοβακία να πω ότι ο ε, Πρωθυπουργό σα επανειλημμένα έχει πει ότι δεν θέλει πρόσφυγες στο εδαφός του. Από την άλλη, πρόσφατα είχαμε Σλοβακική Προεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας είχα πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με τον Ρόμπερτ Κάλνικ, Υπουργό Εσωτερικών. Μετά από πολύ ωραίες ε, συνομιλίες με αυτόν και άλλους υπουργούς από τις χώρες Βίσεκρατ, άρχισα να καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να πάει κανείς από 0 στο 100%, ε, στο 100 της ποσόστοσης ε, εν μία νυχτή. Αυτό είναι δύσκολο να το υπερασπιστεί κανείς απέναντι και στους πολίτες ε, που δεν έχουν συνηθίσει να συναναστρέφονται ανθρώπους από άλλες χώρες. Γι' αυτό στο κείμενό μου ε, προτείνω μεταβατική περίοδο 5 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας ε, προχωράει κανείς από το 0 στο 20% το πρώτο έτος, ε, μετά 40, 60, 80 και φτάνει το 100% μετά από 5 χρόνια. Επίσης, ε, προβλέπουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό και θα πρέπει να έχουμε και κατανόηση απέναντι στα κράτη που ε, έχουν λιγότερες εμπειρίες όσον αφορά την υποδοχή ανθρώπων από άλλες χώρες. εκπρόσωπος ε, της ε, Σλοβακίας ε, μου είπε ότι είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Και νομίζω ότι αν μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε αυτό και άλλα στοιχεία, θα μπορέσει αυτό να γίνει αποδεκτό και από την Τσεχία και από άλλα κράτη-μέλη. Κατόπιν ε, ρωτήσατε αν ε, το Συμβούλιο δεν έχει λέγει. Ε, φυσικά, είμαστε συνομοθέτες. Το Συμβούλιο από τη μία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άλλη και πρέπει να συνεργαστούμε. Και νομίζω ότι στην Ευρώπη σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερη, πολύ περισσότερη συνεργασία. Θα πρέπει να ξεφύγουμε ο καθένας από το δικό του περιορισμένο πεδίο και θα πρέπει να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι να ε, αφήσουμε πίσω μας ε, τους διαθεσμικούς αγώνες που είδαμε στο παρελθόν, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την ε, πραγματική κατάσταση. Ο φίλος από την Τσεχία αναφέρθηκε στο επίπεδο εναρμόνισης. Γνωρίζετε ότι όλες οι προτάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, στοχεύουν σε ένα σύστημα εναρμονισμένο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα που να μην ενθαρρύνει το ίδιο τους ανθρώπους να μεταφερθούν αλλού όπου οι συνθήκες ε, να είναι πιο ευνοϊκές. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς ε, στη βάση και με κάθε λεπτομέρεια, αλλά μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει πρόσβαση ε, στις ίδιες υπηρεσίες, ε, το χρονοδιάγραμμα να είναι λίγο πολύ το ίδιο μεταξύ των κρατών μελών, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κλπ. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για εναρμόνιση. Φυσικά στοιχίζει πιο πολύ να ζει κανείς ε, στη Γερμανία ή στη Σουηδία σε σχέση με ποια χώρα να σας πω, την Τσεχία ίσως. Φυσικά δεν θα πρέπει να λαμβάνει κανείς το ίδιο ποσό σε κάθε χώρα. Θα πρέπει το ποσό αυτό να, αντικατοπτρίζει, να, να αντιστοιχεί στην κατάσταση ε, στο κράτος μέλος αυτό. Το πολύ σημαντικό θέμα, το, ε, το οποίο θα μπορούσαμε να συζητάμε όλη μέρα, ε, είναι η ένταξη στην κοινωνία. Όπως γνωρίζετε, το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην πρόταση αυτή. Είναι θέμα επικουρικότητας. Όμως, Εάν αυτή η νομοθεσία εφαρμοστεί σωστά, θα μπορέσει να καλλιεργήσει ένα, ένα σύστημα όπου να γίνεται σωστά η ένταξη. Δεν είναι σωστό οι άνθρωποι να μην ε, εντάσσονται στην κοινωνία. Ε, πολύ συχνά ε, διάφοροι αναφέρουν την Σουηδία ως καλό παράδειγμα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου καλό. Στην παλιά 7 χρόνια ήταν το μέσο διάστημα για την οικονομική ανεξαρτησία των των μεταναστών που εντάσσονται στην κοινωνία. Τώρα πια όμως είναι εννέα χρόνια. Θα πρέπει να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον, να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Το, το θέμα όμως αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή της νομοθετικής πρότασης που συζητάμε σήμερα. Άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Um, hello, από την Πολωνία επίσης, κυρία Κορπόφσκα. Ένα ερώτημα για τις επιπτώσεις. Ποιε θα είναι οι επιπτώσει ε, εφόσον υπάρχει συμφωνία για τι χώρε που δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το μπουφέ, όπω είπατε, θα υπάρξει κάποια τιμωρία. Θα αλλάξει κάτι στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, θα γίνει κάτι άλλο. Ένα ερώτημα. Μη... Από τη Γαλλία είμαι. Μαγλίν Μπομάρ για τη Μοντ μήπως τελικά θα φτάσουμε σε ένα πολύ ωραίο κείμενο που θα δίνει πολλές εγγυήσεις ε, επιφανειακά και από εκεί πέρα θα υπάρξουν συμφωνίες με χώρες όπως η Τουρκία ε, όπου θα δημιουργήσουμε μια Ευρώπη χωρίς πρόσφυγες, χωρίς τούντες άσυλο με αυτό το, ε, το, το σύστημα με τις μελέτες ε, αποδεκτού ε, με γειτονικές χώρες οι οποίε θα θεωρούνται ασφαλεί και θα πηγαίνουν εκεί οι πρόσφυγε, μήπω τελικά θα φτάσουμε, φτάσουμε μια Ευρώπη χωρί ετούντε άσυλο. Καλό απόγευμα, Μπλά Μωρένο από την Ισπανία. Θέλω να μου πείτε κάτι περισσότερο για το θέμα ε, των ασυνόδευτων ανηλίκων και των φρουρών και των κηδεμόνων τους. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, ε, για εφόσον κάποιος δεν σεβαστεί την νομοθεσία. Ακούστε, την πρόσθεση της Κομισιόν υπάρχει δυνατότητα opt-out. Αλλά αυτό έχει οικονομικές επιπτώσεις. Εάν μια χώρα δεν ε, λάβει, δεν υποδεχθεί πρόσωπα σύμφωνα με το αυτόνομα, αυτόνομος, ε, με το αυτόματο σύστημα κατανομής, στο τέλος του έτους θα γίνει υπολογισμό και 250.000 ε, ε, ανά άτομο θα αφαιρεθούν. Είναι μια οικονομική ύπτωση, ένα πρόστιμο, πέστε το όπως θέλετε. Εγώ αυτό όμως το αφαίρεσα την πρότασή μου. Το θεωρώ μη ηθικό, δηλαδή να βάζουμε μια τιμή στον κάθε άνθρωπο ανακεφάλι. Θέλω όμως να δω πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε πιο αποτελεσματικά. Μιλάμε για ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μιλάμε μόνο για πρόσωπα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορούμε να παρακρατήσουμε ένα μέρος της χρηματοδότησης από τα διευθυντικά ταμεία, τα περιφερειακά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά όντως θα παρακρατούνται στο τέλος του έτους εφόσον κάποιος δεν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να, το, να εξεταστεί περαιτέρω. Στην Περιφερειακή Επιτροπή υπήρξαν κάποιες τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ε, η αντίληψη και στο Συμβούλιο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Όλο και περισσότεροι υπουργοί ε, γράφουν άρθρα, λένε δημοσίως ότι του αρέσει αυτή η ιδέα, θέλουν να συμβεί αυτό. Και υπάρχει μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Να υπάρχει δηλαδή κάποια οικονομική επίπτωση, εφόσον κάποιο δεν συμμορφώνεται, εφόσον κάποιο δεν αναλαμβάνει το μέρο τη ευθύνη που τον αλογεί. Τώρα, κάποιες χώρες, μια από τις χώρες είναι και η δική σας, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γίνεται αντιληπτή ως οικονομική αλληλεγγύη. Μου λένε δηλαδή, εάν παρακρατήσετε χρήματα, αυτό είναι κατά της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Προς αυτές τις τέσσερις χώρες, αλλά και άλλες ενδεχομένως, εγώ θα έλεγα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει ότι είμαστε, λένε, είμαστε χώρες οι οποίες λαμβάνουν χρήματα από δέκτες και αυτό πρέπει να συμβεί διότι αυτό το σύστημα των διαθροτικών ταμείων έχει ως στόχο να μειωθεί η απόκληση μεταξύ των φτωχών και των πλούσιων χωρών. Αν μιλήσετε δηλαδή με έναν απλό πολίτη στις χώρες αυτές, αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει ενδεχομένως. Στη χώρα μου όμως και σε άλλες 20 χώρες, μπορεί και παραπάνω. Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι η κάθε χώρα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της έχουμε μια κοινή δέσμευση. Η κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να λάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Αυτό είναι η αλληλεγγύη. Ό, όταν μιλάω εγώ στους γειτονές μου, στη γειτονιά μου. Μπορεί εσείς όταν μιλάτε στους γειτονές σας να η να είναι, ε, είναι θέμα χρημάτων. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά αντίληψης. Νομίζω ότι και τα δύο μπορούν να γίνουν. εφόσον συμμορφωθούμε με την νομοθεσία δημιουργούμε αλληλεγγύη και προχωράμε. Δεν είναι όμως βιώσιμο πλέον οι πέντε χώρες που λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα. Δεν μπορεί να, γίνει, να κάνουν κάποιοι το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας και κάποιοι να κάνουν πολύ λίγη προσπάθεια ή καθόλου. Τώρα, για την εξω... Ε, το, το, να, δημιουργούμε τρίτες χώρες, ε, να αναλαμβάνουν τρίτες χώρες την ευθύνη, ε, αντί για μας και ουσιαστικά να διαβρύνουμε τα εξωτερικά σύνορά μας. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δείχνει, κατ' εμέ, ακριβώς αυτό. Βεβαίω υπήρξε αυτή η συμφωνία διότι έπρεπε κάτι να γίνει εκείνη τη στιγμή εφόσον δεν λειτουργούσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Το ίδιο ισχύει και με τα 160 άτομα τα οποία πρέπει να ε, μετακατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα. Είναι θέμα λειτουργίας του συστήματος ασύλου. Παίρνουμε αυτά τα μέτρα, τα επίγοντα, κλείνουμε σύνορα. Το 2015 συνέβη αυτά. Ε, διακυβεύθηκε ο χώρος έγκεν. Και πάλι αυτό ήταν ένα μέτρο κατεπήγον επειδή λειτουργεί το σύστημα. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτή τη στιγμή να θεσπιστεί ένα σύστημα το οποίο να εγγυάται ότι ο χώρος Σέγγεν θα διαφυλαχθεί. Ένα σύστημα όπου θα μοιραζόμαστε την ευθύνη, θα συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις αυτές. Και βεβαίως ε, αναφερθήκατε και στην αρχική ε, αξιολόγηση σχετικά με τον έννοια της ασφαλούς χώρας. Βεβαίως κάποιες χώρες είναι πιο ασφαλείς από άλλες. Όμως πάντα μπορεί κάποιος, ένα πρόσωπο, να μην θεωρείται ότι μπορεί να είναι ασφαλής σε μία χώρα. Πρέπει δηλαδή το αίτημα ασύλου να εξετάζεται σύμφωνα με συνθήκη της Γενέβης, σύμφωνα με τη ε, διεθνή νομοθεσία αλλά και την ευρωπαϊκή. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει τα ιστορικά μας σύνορα να τα αναθέσουμε σε άλλους. Πρέπει να λάβουμε εμείς την ευθύνη. Να σας πω μια ιστορία. Εγώ εκπροσωπούσα το Κοινοβούλιο στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής για το άσυλο και μετανάστευση στη Νέα Υόρκη πέρυσι. Για πρώτη φορά. Και αυτό οδήγησε στη δήλωση της Νέας Υόρκης για τη μετανάστευση. Διαβάστε την, είναι ενδιαφέρουσα. Είναι διαφορετική από τα ευρωπαϊκά έγγραφα. Και εκεί αναφέρεται σαφώς σε αυτήν την συνάντηση υψηλού επίπεδου ότι 85% των ετούντων άσυλο στον κόσμο αφορούν αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που έχει να κάνει με την Ευρώπη και που φτάνει στην Ευρώπη. Ακόμα και το 2015 όταν υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι μας πλημμυρίζουν, ακόμα και τότε 0,2% του πληθυσμού μας ε, ε, ε, προσωπούσαν αυτοί οι πρόσφυγες. Ο Λίβανος είναι μια χώρα 4,5 εκατομμυρίων. Ένα στους τέσσερις ανθρώπους εκεί είναι πρόσφυγας. 25-30% του πληθυσμού. 0,2 εμείς στην Ευρώπη. Συγκρίνετε το. κάνετε τις συγκρίσεις. Στην ίδια διάσκεψη στη Νέα Υόρκη συνάντησα έναν ε, υπουργό από την Αιθιοπία ο οποίος μου είπε εντάξει ε, είστε η πιο πλούσια περιοχή του κόσμου και δεχτήκατε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπου σε ένα χρόνο. 28 χώρε είσαστε έτσι. Στη χώρα μου ορισμένε φορέ έρχονται 3-4 εκατομμύρια όταν λαμβάνει η χώρα κάποια καταστροφή κάπου κοντά μα. Πρέπει αυτόν να το αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ε, τα μεγέθη. Είμαστε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και να δούμε πώς θα συνεργαστούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κηδεμόνες, για τους ε, τους ανηλίκους, πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες έτσι ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ποτέ να μην κινδυνέψουν να γίνουν προϊόν εκμετάλλευσης ε, ή να μην καλυφθούν οι ανάγκες τους. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και το να καθορίσουμε και δαιμόνες, αυτό να ορίσουμε δαιμόνες είναι κάτι που ζητούν ομόφωνα όλες οι ΜΚΟ οι οποίες εργάζονται στον τομέα αυτών. Πρέπει να ολοκληρώσουμε νομίζω. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ σαφή όλα αυτά. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος του προγραμματός μας όπου έχουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Όπως εξήγησα πριν, όταν μίλησε ο Ρίκε, η διαδικασία στο Κοινοβούλιο έχει ως εξή. Υπάρχει ένας εισηγητής, σε αυτή την περίπτωση η κυρία Βέξτρομ, και μετά κάθε πολιτική ομάδα ορίζει έναν βουλευτή ή μια βουλευτή που αναλαμβάνει το θέμα για να τον απτύξει από τη δική του άποψη από την άψη της ομάδας του. Στο πάνελ λοιπόν μαζί μου για αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Ε, ε, έχω τη χαρά να καλωσορίζω τον κύριο Γιούση Χαλαάχο από την ομάδα ECR ε, στη Φιλανδία, την κυρία Αλεσάνδρα Μουσολίνη από το ΕΛΚΑ στην Ιταλία, από την Ιταλία, συγγνώμη, την κυρία Τζιν Λάμπερτ από την ομάδα των Πρασίνων και από το Ενωμένο Βασίλειο. Επίσης θα έχουμε την κυρία Έλλη Σλάιν από τους Σοσιαλιστές, και την κυρία Λάουρα Φεράρα από την ομάδα EFTD, αλλά οι δύο αυτές τελευταίες ομιλήτρες θα καθυστερήσουν λίγο. Okay. I, please, please try and be quiet. If you're going exit the room, please keep... Παρακαλώ, αν φεύγετε από την αίθουσα, αποχωρείτε ησύχως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Με ποιον να ξεκινήσουμε. Είναι κάποιο που πρέπει να φύγει νωρίτερα, ο κύριο Χαλάου, ίσως. Ωραία, ευχαριστώ. I, I think what's really interesting to... Αυτό που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ε, για τους δημοσιογράφους εδώ και που θα ήθελα να καταλάβουν να τους εξηγήσετε τις θέσεις των ομάδων σας. Τι πιστεύει δηλαδή η ομάδα σας για το θέμα αυτό. Ε, η συγγήτρια ανέφερε καθαρά τις διάφορε συμβιβαστικές, τους διάφορου συμβιβασμούς. Πρέπει να μας δείξετε, δηλαδή να μας πείτε σε ποια σημεία υπάρχει κάποιο επίπεδο συμφωνίας, που υπάρχει διαφωνία για τα διάφορα σημεία αυτού του θέματος. Σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Εκπροσωπώ τον συνάδελφό μου, Ντάνιελ Ντάλτον, που είναι ο ε, σκιώδης εισηγητής ε, για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Ο Ντάνιελ ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα, θα κάνω όμω κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσεις εκ μέρου του και στο όνομα της ομάδας μας. Δυστυχώ, και εγώ δεν θα μπορέσω να παραμείνω για όλη τη συζήτηση, διότι έχω ανηλυμένε υποχρεώσει. Η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου εξ αρχής ήταν θέμα δύσκολο με ελάχιστη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο λόγος που απέτυχε ε, το σύστημα κατά την ε, μεταναστευτική κρίση δεν ήταν μόνο ότι ήταν ελαττωματικό το σύστημα, ήταν και ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, τήρησαν τις υποχρεώσεις τους και η συνεργασία έφτασε πολύ αργά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αναθεώρηση αυτή να έχουμε κατά νου την εφαρμογή του κανονισμού στα κράτη-μέλη και να προωθήσουμε ένα σύστημα το, με το οποίο να μπορούν να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης αλλά και μακροπρόθεσμα. Αυτό δεν σημαίνει κυρώσεις στα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται ή να, βάλουμε, να ορίσουμε τιμή για τον κάθε πρόσφυγα, για να επιβάλλουμε πρόστιμο στα κράτη-μέλη για κάθε ε, πρόσφυγα που δεν ε, υποδέχονται. Θα πρέπει λοιπόν ε, το, να ξαναποκτήσουμε τον έλεγχο του συστήματος, δηλαδή να μειώσουμε την εισρωή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο αν αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές αιτίες της κρίσης με έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, με σωστή καταχώρηση καθενός που καταφτάνει στα ε, σύνορα και διασφαλίζοντας ε, σωστές επιστροφές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ξαναδημιουργήσει εμπιστοσύνη στο σύστημα και να θα έχει το δυναμικό ώστε να δώσει στους πιο ευάλωτους ε, ετούντες άσυλο ε, τα μέσα που είναι απαραίτητα. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και εναρμόνιση για να αποθαρρύνουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις ε, και την αναζήτηση του ευνοϊκότερου καθεστώτος ασύλου εντός της Ευρώπης από πλευράς των ετούντων. Οι διαδικασίες όμως θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην κάνουν πιο ελκυστική την Ευρώπη στα μάτια αυτών που χρησιμοποιούν τη διαδικασία ασύλου ως τρόπο οικονομικής μετανάστευσης. Εγκαταλείποντας την αρχή της πρώτης χώρας εισόδου, μπορεί να καταλήξουμε σε τέτοια ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Η κυρία Μουσολίνη, στο όνομα του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα Ιταλικά γιατί είναι προτιμότερο. Εμείς ε, με αυτό τον νέο κανονισμό θέλουμε και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συμφωνούμε με την εισηγήτρια σε πολλά θέματα πέραν ε, των ε, διαφορετικών απόψεων και κάποιων πτυχών. Θέλουμε να είμαστε πολύ θαραλέοι και φιλόδοξοι. Η κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι τρομακτική από όλες τις απόψεις. Ανθρωπιστικά και από άποψη ασφάλειας. Εξακολουθούν να καταφτάνουν σκάφη γεμάτα ανθρώπους. Στην Ιταλία, όπως ξέρετε, γράφτηκαν κάποια πράγματα για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, που μεταφέρουν, όπως λέγεται, μετανάστες ε, στην Ιταλία κυρίως και που αντί να φτάνουν στο κανάλι της Ικελίας ε, μεταφέρονται κατευθείαν στην Ιταλία. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η αναθεώρηση του Δουβλίνου. Γιατί, διότι πολλοί μετανάστες δεν θέλουν να ενταχθούν στον κανονισμό του Δουβλίνου, διότι δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ιταλία. Εμείς λοιπόν αντιμετωπίσαμε το εξή πρόβλημα. Δεν ήθελαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία δεν είναι καν υποχρεωτικά. Ουσιαστικά Θέλουμε, ε, και αυτό φαίνεται ουτοπικό φυσικά ε, ειδικότερα τώρα, θέλουμε να κάνουμε πιο δημοφιλή την αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη. Δηλαδή να καταφέρουν και οι άλλοι όπως η Ιταλία να υποδεχθούν ε, τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και από τις διώξεις. Κάτι άλλο που θέλουμε να κάνουμε στο πλαίσιο ενός άλλου κανονισμού όπου η δική μας θέση του ΕΛΚ αντιτίθεται κάθετα ε, στη θέση της εισηγήτριας για τις ελάχιστες απαιτήσει, δηλαδή τον κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσει, δηλαδή για το ποιος έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στην διεθνή ε, προστασία ως ε, πρόσφυγας ή στο πλαίσιο της επικουρικής προστασίας, διότι θέλουν να επεκτείνουν και στους ε, κλιματικούς ας πούμε μετανάστες, τους μετανάστες για λόγους κλιματικών αλλαγής, ε, στο, το οποίο μας βρίσκει αντίθετους. Και το θέμα της οικογένειας ε, που έχει δημιουργηθεί μετά από την άφηξη. Θέλω να ενταχθεί και η οικογένεια που έχει δημιουργηθεί μετά την άφηξη του μετανάστη στο επικράτεια των κρατών μελών. Αυτά είναι δύο θέματα για μας πολύ ευαίσθητα, μας δημιουργούν πρόβλημα στο ΕΛΚΑ και είμαστε κατά. Διότι αυτό θα αποτελούσε παράγοντα έλξης, τεράστιο μάλιστα, φανταστείτε. Ε, στο Δουβλίνο, με αυτό το αυτοματοποιημένο δίκτυο που εισάγει η Κομισιόν και που επέκτηνε η κυρία Βίξτρομ, εμείς ε, συμφωνούμε. Διότι να διανομήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια πέρα των χωρών που θα έχουν κάποια μεταβατική περίοδο γιατί δεν έχουν συνηθίσει. Ε, όπως λένε. Ε, ναι, νομίζετε ότι συνηθίζει ποτέ κανείς, τέλος πάντων. Και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συνηθίσουν και να προσαρμοστούν. Ε, εμείς λοιπόν ε, αντιτιθέμεθα σε διάφορες τροπολογίες με κάποιες συνεργασίες παρότι με τους, με τους σοσιαλιστές, με τους πράσινους, με βλέπουμε κάποια θετική εξέλιξη με τον άλλο κανονισμό καθόλου. Ο άλλος κανονισμός δημιουργεί πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μετά. Ας ακούσουμε την κυρία Τζιν Λάμπερτ πρώτα, εκ μέρους των Πρασίνων. Ποια είναι η θέση της ομάδας των Πρασίνων για το θέμα αυτό του κοινού συστήματος ασύλου. Θα μπορούσατε να το συνδέσετε επίσης ε, και με τη γενικότερη θέση σας και για τις υπόλοιπες οδηγίες. Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να βρίσκομαι εδώ. Σε ό,τι αφορά το Δουβλίνο, δεν θα σας εκπλήξει αν σας πω ότι οι πράσινοι ποτέ δεν ήταν ε, θερμοί υποστηρικτέ του συστήματος του Δουβλίνου, του κανονισμού του Δουβλίνου όπως, λειτουργεί ως τώρα. Πέρσι εργαστήκαμε ως πολιτική ομάδα προσπαθώντας ε, ε, να δούμε ποια θα είναι η εναλλακτική στο Δουβλίνο 1, 2 ή 3. Όταν βλέπουμε τις προτάσεις τώρα που βρίσκονται επιτάπητος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την εισηγήτρια την κυρία Βίξτρομ, η θέση μας ε, βεβαίως πάντα πηγάζει από το δικό μας έγγραφο. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει ένα σημείο όπου συμφωνούμε με το ECR. Ε, το παρόν σύστημα αυτή τη στιγμή είναι ε, αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες δεν πετυχαίνει το βασικό σκοπό δηλαδή η σε και δίκαιη αξιολόγηση ενός αιτήματο ασύλου δεν είναι βέβαια μόνο αυτό ε, εμείς λοιπόν καταρχήν είναι σαφές ότι το Δουβλίνο δεν λειτουργεί για μας σε ό,τι αφορά ε, την οικογενειακή επανένωση, ό,τι αφορά του ασυνόδου ανηλίκου. Ε, εγώ είμαι το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό που συμβαίνει μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλία, παραδείγματο χάρη, ε, είναι τραγικό. Θέλουμε λοιπόν ένα σύστημα που να λειτουργεί καλύτερα και για τα κράτη-μέλη και για του εντούτε άσυλο και τα προβλήματα που θέλουμε να επιληθούν έχουν να κάνουν με το πώ θα απομακρυνθούμε από αυτή τη συγκέντρωση σε κάποιε χώρε έχουμε δει ότι αυτό αφορά η Ισπανία, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία ενδεχομένω, ανάλογα και με την κατάσταση στην Ουκρανία, η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ετούντες άσυλο που δεν καταγράφονται, οι πιο ευάλωτοι χάνονται, έχουμε όλο και πιο πολλούς, πιο πολλούς παράτυπους μετανάστες. Ε, οι δευτεραγενείς μετακινήσεις και γιατί συμβαίνει αυτό και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την, την αίσθηση αταξίας που υπάρχει από το 2015. Και κάθε χώρα το προσεγγίζει το θέμα με βάση τη δική της λογική. Ε, εμείς θέλουμε να απομακρυνθούμε από τις καταστάσεις εκείνες όπου η ο ετών άσυλο έχει μόνο μία ευκαιρία και αυτή η ευκαιρία πικίλια προς ποια χώρα απευθύνεται ε, το πώς η κάθε χώρα ερμηνεύει και εφαρμόζει το κεκτημένο περί ασύλου. Όταν έχει λοιπόν κάποιος μόνο μία ευκαιρία και παγιδευτεί σε μία χώρα θα πρέπει να μείνει εκεί για όσο έχει άδεια παραμονής τότε ναι, οι άνθρωποι θα νιώσουν παγιδευμένοι και θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε αυτή η μία ευκαιρία που έχουν να, έχει, να έχει όσο γίνεται περισσότερε πιθανότητε να πετύχει. Αυτά σκεφτήκαμε όταν υποβάλαμε τη δική μα πρόταση που υπάρχει στην ιστοσελίδα μα. Έχει να κάνει λοιπόν με το να, να, να μοιραστεί η ευθύνη στα κράτη-μέλη. Δηλαδή να ε, μειωθεί η πίεση προς κάποιες χώρες ε, να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Ήταν σημαντικό να αποσυρθεί η πρόταση της πρώτης χώρας εισόδου, ε, όπως κάνει και η συγγήτρια, το γεγονός ότι εξετάζουμε ε, τους ε, πρόσφυγες ως κοινότητες, ότι θα πρέπει να γίνουν ομαδικές κατανομές. να μην υπάρχει βεβαίω απόλυτη ελεύθερη επιλογή για του ετούντε άσυλο, αλλά να έχουν κάποιες επιλογέ. Έτσι λοιπόν ε, δεν πρέπει η πρώτη χώρα εισόδου, το πρώτο, η πρώτη επαφή να καθορίζει το μέλλον. Μπορεί κάποιος ε, να έχει ήδη κάποιους δεσμούς με κάποια χώρα ε, και αυτό να του δίνει την δυνατότητα να κάνει κάποια επιλογή. Πρέπει να υπάρχει αυτό κατά μας. Είναι σημαντικό. Γίνονται συζητήσει σε επίπεδο πολιτικών ομάδων που πάνε προ σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια που θα καταλήξουν. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα κινείται προς την κατεύθυνση ε, που εμείς θα προτιμούσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι παρότι υπάρχουν διαφορές τις οποίες ε, σαφώς αναφέρατε σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Βίξτρομ προηγουμένως. Ε, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και κάποια σημεία σύγκλησης, τουλάχιστον επί τη βάση της ανάγκης μεταρρύθμισης του συστήματος, ε, της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών, το θέμα της καταγραφής, ε, της εγγραφής και των δευτερογενών ε, μετακινήσεων, αυτά φαίνεται να είναι σημεία σύγκλησης. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξει συμφωνία ή πιστεύετε ότι τελικά θα έχουμε ένα αποτέλεσμα κάπως νερωμένο. Ας δούμε το κείμενο. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι για το Δουβλίνο θα βρούμε συμφωνία, διότι υπάρχει σύγκληση επί των σημαντικών σημείων. Θα πρέπει τώρα να δούμε τι θα συμβεί και στο Συμβούλιο. Προσοχή διότι εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε κάποια συνοχή απόψεων, αξιολογούμε, συζητάμε. Αν όμως το κείμενο αποτελέσει το αντικείμενο αρνησικήριας ή αλλαγών σημαντικών στο Συμβούλιο, δεν ξέρω τι θα συμβεί, μην το ξεχνάμε. Εγώ ελπίζω ότι το Συμβούλιο δεν θα πάει και να πει «Α, μπλοκάρουμε τα πάντα γιατί θέλουμε το παλιό κείμενο», το οποίο σημαίνει ότι εκεί το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία σημασία. Αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό. Κύριε Λάμπερτ. Yeah, I think that, you know... Ένα από τα πράγματα που θα δούμε, όπως είπε και η συνάδελφος, είναι ότι το, ότι το Συμβούλιο όπως ε, πολύ συχνά θα θεωρούσε κανείς, θα αποτελέσει μέρος του προβλήματος. Χρειάζεται αλληλεγγύη και το είδαμε αυτό και στις διασώσεις στη θάλασσα και στον τρόπο που λειτουργεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Χρειάζεται τα άλλα κράτη-μέλη να βοηθήσουν ε, αυτά που βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση. Νομίζω ότι βλέπουμε κάποιες εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες... Και προσπαθώ να βρω, να βρω τρόπο να το πω ευγενικά, που δεν συνεργάζονται επικοδομητικά. Η συνθήκη μας δεσμεύει να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Ε, κάποια κράτη-μέλη λοιπόν θέλουν να επιδείξουν αλληλεγγύη με το δικό τους τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να επιστρέφουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα εισόδου. Νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρχίσει να επιστρέφει περισσότερο στη Γερμανία. Επανερχόμαστε λοιπόν στην κατάσταση όπου δεν ε, εξετάζουμε τις αιτήσει ασύλου, Φαίνεται σαν κάποια κράτη-μέλη να μην θέλουν να ε, ε, να είναι διατεθειμένα να κάνουν οτιδήποτε, αρκεί να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτό δεν βοηθά ούτε τη διεθνή μας φήμη, ούτε βοηθάει τις εσωτερικές εργασιακές σχέσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο για να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ και πάλι, σηκώστε το χέρι σα. Μπορείτε να θέσετε τι ερωτήσεις σας όχι μόνο στα αγγλικά, αλλά και στις ε, γλώσσε που παρέχετε διερμηνία. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ. My name is Catherine. Το όνομα είναι Κάθρι Μέρκαλη από, την Φιλανδία, συγγνώμη. Ένα ερώτημα προ την κυρία Λάμπερ. Αναφερθήκατε στο ζήτημα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά επί ποιας βάσης χορηγούν άσυλο για έναν ετών άσυλο από το Ιράκ. Οι πιθανότητες του ε, να πάρει άσυλο στη Φιλανδία ε, είναι πολύ χαμηλότερες από ότι να ε, δεχτεί άσυλο, να, να, να, του χορηγηθεί το άσυλο στη Γερμανία. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητείται πολύ. Πώς σκοπεύετε να το εντοπίσετε. Ναι, είναι αλήθεια. Ο κανονισμός του Δουβλίνου βέβαια δεν ασχολείται ακριβώς με αυτό, αλλά ε, στον παρόν κανονισμό, στις τελευταίες διαπραγματεύσεις έγινε μια πρόταση από την Πολωνική Προεδρία έτσι ώστε τουλάχιστον να κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να γίνεται και μια αξιολόγηση ομοτήμων από χώρα σε χώρα ε, δηλαδή ε, ειδικοί που εργάζονται στα πλαίσια του ΕΑΣΟ να εξετάσουν από κάθε χώρα κατά πόσο ε, λειτουργούν σωστά τα συστήματα. Ε, ήταν βέβαια δύσκολη η συζήτηση για το θέμα αυτό. Οι χώρε ε, δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα, τα κράτη-μέλη, δηλαδή ότι κάποιο θα να του πει κατά πόσο το σύστημά του είναι καλό ή όχι και κατά πόσο λειτουργεί. Ήταν ένα σημαντικό βήμα στα πλαίσια του Δουβλίνου 3. Βεβαίω υπάρχει ε, το θέμα ότι η οχι κατα ποσο λειτουργει ηταν ενα σημαντικο βημα στα πλαισια του δουβλινου 3 βεβαιω υπαρχει το θεμα οτι η ασο θα γίνει υπηρεσία, θα γίνει οργανισμό, δηλαδή κανονισμό, κανονικό. Οπότε θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για το πώ λειτουργούν τα σύστημά του, η ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων, υπάρχει, υπάρχουν κάποιε κατευθύνσει γραμμέ ε, για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Η χώρα προέλευση και σχετική πληροφορία ε, που είναι όλο και πιο σημαντική όταν δείτε τα ποσοστά αποδοχή ε, και χορήγηση ασύλου για χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αυτό ήταν μέρος της λογικής. Λοιπόν, να υπάρξει αυτή η υπηρεσία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ενημερώνονται για το τι γίνεται αλλού και να υπάρχει μια ευθυγράμμιση σιγά-σιγά. Αυτό είναι ένα εξελίξη. Όταν βεβαίως βλέπουμε τι γίνεται με το Δουβλίνο, ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους όταν κάποιος κάνει μια αίτηση ασύλου και βρίσκεται σε μια χώρα όπου είναι πολύ, ε, πολύ λίγε πιθανότητε να λάβει κάποιο άσυλο, στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, 1% πριν από μερικά χρόνια ήταν ε, το ποσοστό. Ή ε, γνωρίζει κάποιο ότι υπάρχουν διαφορέ. Ε, δεν προκαλεί έκπληξη ότι αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνται. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο ζητούμε εδώ και καιρό από τα κράτη-μέλη να υπάρξει ευθυγράμμιση των συστημάτων. Ε, και αυτό έχει να κάνει με τη εργασία της ε, ε, υπηρεσίας υποστήριξης ασύλου που θα έχει τις απαραίτητες ε, ε, δεξιότητες για να το κάνει αυτό. Όλα αυτά βρίσκονται που επανεξέταση αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Στο πάνελ τώρα έρχονται δύο ακόμα ευρωβουλευτές από δύο ακόμα πολιτικές ομάδες. Η Έλλη Σλάιν εκπροσωπεί τους σοσιαλιστές και δημοκράτες από την Ιταλία και η Λάουρα Φεράρα εδώ δεξιά μου που, εκπροσωπεί, που είναι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα EFDD από την Ιταλία πάλι. Έχουμε λοιπόν εδώ πλειοψηφία Ιταλών. Ιταλίδων πιο συγκεκριμένα. Ακούσαμε την κυρία Λάμπερ, την κυρία Μουσολίνη και είδαμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης σε ό,τι αφορά τις θέσεις των πολιτικών ομάδων για το θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως και αποκλήσεις. Θα ήθελα τώρα η κυρία Σλάν και η κυρία Φεράρα ενδεχομένως ε, να μας παρουσιάσουν ποια είναι η θέση των πολιτικών τους ομάδων για το θέμα. Βεβαίως μπορείτε να μιλήσετε ιταλικά εφόσον το επιθυμείτε, διερμηνία υπάρχει. Όπως θέλετε. Ε, μιλήσω αγγλικά, ευχαριστώ μπορεί αυτό να είναι ευκολότερο για εσά για να με καταλάβετε. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Άργησε το αεροπλάνο που με έφερε εδώ κατά μία ώρα. Η θέση της ομάδας μας. Εδώ έχουμε μια ωρα η θεση τη ομαδα μας εδω εχουμε μια ευκαιρια επιτελου ε, να ξεπεράσουμε αυτό που ονομάζω εγώ την αρχική υποκρισία του συστήματος του Δουβλίνου. Δηλαδή ότι το Δουβλίνο επιβάλλοντας αυτό το κριτήριο της πρώτης χώρας παράτυπης εισόδου που ε, υποτίθεται ήταν το τελευταίο κριτήριο το, ήταν το άρθρο 15 του κανονισμού τελικά κατέληξε να είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω οπότε μέσα στα χρόνια σε αυτό οφειλόταν στο μεγαλύτερο βαθμό ε, τα αιτήματα ασύλου ε, στα κράτη-μέλη που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Οπότε η πρότασή μας βασίστηκε σε μια απλή αρχή. Όποιος ξεφεύγει από πόλεμο ή δίωξη δεν πάει σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει την ευθύνη και να τους καταμερίσει ίσα, ισότιμα. Δεν λέμε να επινοήσουμε κάτι καινούριο διότι οι συνθήκες ήδη μας το απαιτούν στα άρθρα 78 και 80 που αναφέρονται σε αλληλεγγύη και ίση κατανομή των ευθυνών. Αν δούμε τα στοιχεία των τελευταίων ετών, βλέπουμε ότι 6 κράτη-μέλη από τα 28 αντιμετώπισαν το 80% όλων των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αλληλεγγύη, αυτή είναι ίση κατανομή των ευθυνών, ε, όπως ε, διέπονται και προβλέπονται από τις συνθήκες. Δεν νομίζω. Κάτι άλλο που ζητάμε είναι να υπάρχει κάποια συνοχή με κάτι που έχει ήδη ψηφίσει πάνω από μία φορά στο Κοινοβούλιο αυτό, διότι πάνω από μία φορές ε, στο Κοινοβούλιο το παρόν έχουμε ψηφίσει την κοινή ευρωπαϊκή λύση που χρειαζόμαστε απελπισμένα γιατί είναι σαφές για όλους ότι η μετανάστευση και το άσυλο είναι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του. Για να υπάρχει λοιπόν ε, συνοχή με το ψήφισμα Κέγγε Μετσόλα που πέρασε πέρσι τον Απρίλιο όπου ζητήσαμε να παραβλέπετε το κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου και να κινηθούμε προς μια συγκέντρωση των ευθυνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το άσυλο η βασική αρχή είναι κάτι που μας αρέσει να συζητάμε όταν πάμε σε άλλα κράτη-μέλη. Και μιλώντα και για το Συμβούλιο, ξέρει ότι αναφέρθηκε σε αυτό η Τζιν πριν έρθω, είναι ντροπή. Ντροπή. Όχι μόνο που δεν κατάφεραν ε, να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις σε θέματα μετεγκατάστασης, τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το Σεπτέμβριο του 2015. Μην ξεχνάμε ότι ε, ε, υπελείπεται 11-12% της ε, συνολικής δέσμευσης και είναι ντροπή. Πέρυσι στη Νέα Υόρκη, στην πρώτη σύνοδο κορυφής για τους μετανάστες και πρόσφυγες στα Ηνωμένα Έθνη, συζητήσαμε όλα αυτά και ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των το μεγαλύτερο κομμάτι μάλλον των προσφύγων στον κόσμο φιλοξενούνται από αναπτυσσόμενες χώρες, όχι από εμά και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πώ θα αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης όταν όλες οι πολιτικές του Συμβουλίου και τελευταία δυστυχώ και τη Κομισιόν όπω φαίνεται κινούνται κατά κάποιο τρόπο προς την εξωτερική ανάθεση των ευθυνών μας και των συνόρων μας σε άλλου. Δεν είναι σωστό αυτό. Κάθε προσπάθεια εφόσον κατανεμηθεί ισότιμα ε, θα είναι βιώσιμη για όλους. Στην πρότασή μα εμεί έχουμε υποβάλει 145 τροπολογίε. έχουμε συνεργαστεί στενά με τις άλλες ομάδες και προσπαθούμε να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένα άλλο Δουβλίνο που να μην βασίζεται στο ε, άδικο κριτήριο της πρώτης χώρας εισόδου και να βασίζεται σε εύκολα, εύκολα εφαρμόσιμα κριτήρια και σε έναν μηχανισμό μετεγκατάστασης μόνιμο και συγκεντρωμένο, χωρίς κατόφλια χωρίς όρια, διότι το σκεπτικό εδώ είναι ότι όλη η Ένωση είναι ευθύνη για οποιαδήποτε αίτηση ασύλου υποβάλλεται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Οπότε το θέμα είναι πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό. Πρώτα, αρνούμαστε την τιμωρητική προσέγγιση της Κομισιόν, την αντικαθιστούμε με κάτι που εμεί θεωρούμε πιο αποτελεσματικό, να υπάρχουν κίνητρα συμμόρφωσης με το σύστημα και αποθάρρυνση των δευτερογενών μετακινήσεων. Για να τι αποθαρρύνουμε αυτέ τι δευτερογενείς μετακινήσεις πρέπει να δούμε τι αιτίε του. Εγώ βρισκόμουν στο κόμμα, στα σύνορα μεταξύ Ιταλία και Ελβετία φέτο το καλοκαίρι. 500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 200 ανηλίκων, κοιμώντουσαν στους δρόμου. Γιατί? Διότι δεν ήθελαν να ζητήσουν άσυλο στην Ιταλία, διότι ξέρουν τον κανονισμό του Δουβλίνου καλύτερα από εμά. Και δεν ήθελαν να κολλήσουν σε μία χώρα για δύο χρόνια, περιμένοντα μια πολύ απλή οικογενειακή επανένωση με τη μητέρα τους, με το θείο τους σε ένα άλλο κρατό μέλος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούν αυτοί να πληρώνουν τη δική μας ανικανότητα να τους παρέχουμε ένα καλύτερο, πιο αποτελεσματικό σύστημα. Το θέμα μας λοιπόν είναι το εξής, για να είμαι σύντομη. Διαγράφουμε τους ελέγχους ε, παραδεκτού που λέει η Κομισιόν θεωρούμε ότι είναι λάθος, βασίζονται σε ασαφείς έννοιες ε, της ασφαλούς τρίτης χώρας, Θυμάστε κάτι πέρυσι έγινε με την Τουρκία. Το ίδιο συμβαίνει και με μερικέ αφρικανικέ χώρε με το νέο πλαίσιο εταιρική σχέση και τώρα συζητούν και με τη Λιβύη, η οποία δεν έχει καν υπογράψει τη σύμβαση τη Γενέβη. Για μας λοιπόν αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Επίσης στις τροπολογίε μα ενισχύουμε τη διάταξη ενημέρωση, την προβλήση ενημέρωση. σε συμφωνία με τα όσα προτείνει η κυρία Βουέξτρομ, ε, ενίσχυση των δικαιωμάτων των ετούντων και έχει αγκαία για τους ανήλικους ε, και τον αναλαμβάνεται υπόψη το συμφέρον τους ε, με τη σχετική αξιολογία. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα προτείνουμε καταγραφή στην πρώτη χώρα. Ενδιαφέρει όλε τι αρχέ όλων των κρατών μελών να γνωρίζουν ποιο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα αν είναι ευάλωτοι. Και μετά η εύκολη διαδικασία οικογενειακή επανένωση όπω προτείνει η κυρία Βίξτρομ είναι εξαιρετική ιδέα. Ένα από του λόγου που κάποιοι ε, πραγματοποιούν δευτερογενεί μετακινήσει είναι διότι ε, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο οι διαδικασίε. Οπότε η διαδικασία αυτή ε, διευρύνει την πολύ περιοριστική έννοια τη οικογένεια όπω έχει σήμερα στον κανονισμό. Σήμερα, ξέρετε, για παράδειγμα, είναι αδύνατο να επανενωθεί κανεί με μέλο οικογένεια που δεν είναι ετών πρόσφυγα ή ετών άσυλο Εμεί ζητάμε δηλαδή απλά να μπορεί κάποιο να επανενωθεί με ένα συγγενή του που διαμένει νόμιμα σε ένα άλλο κράτο μέλο. Και θέλουμε και τα ενήλικα παιδιά. Ένα γιο άνω των 18 να μπορεί να επανενωθεί με τη μητέρα του. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στον κανονισμό και εμεί θέλουμε να υπάρχει. Και μετά από αυτή την εύκολη οικογενειακή διαδικασία θέλουμε πολύ γρήγορα να ελέγχονται και τα υπόλοιπα κριτήρια του Δουβλίνου στην πρώτη χώρα για να δουν, βλέπει κανείς αν ισχύουν και εμείς προτείνουμε και μια χορηγία, δηλαδή ένας οργανισμός που ε, θα πληρεί κάποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να φιλοξενεί τους ετούντες μέχρι να ολοκληρωθεί η διεκπαιρέωση της αίτησής τους. Και μετά, αν δεν ισχύει κανένα από όλα αυτά τα κριτήρια, θα πρέπει να υπάρχει άμεσα ένας μηχανισμός μετακατάστασης προς ένα άλλο κράτος μέλος που θα λαμβάνει υπόψη τις ε, σχέσεις ε, που έχει ενδεχομένως ο ετών με το κρατός αυτό. Αυτή είναι η δική μας πρόταση και άλλων ομάδων πρόταση είναι. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Και τέλος, αν δεν υπάρχει κάποια σχέση ε, του ετούντο με μια χώρα, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης ο ετών θα πρέπει να έχει κάποια επιλογή, κάποια δυνατότητα επιλογής μεταξύ, για παράδειγμα, των έξι κρατών μελών που δεν έχουν ε, ε, καλύψει την ποσόστοση που αντιστοιχεί σε κάθε κρατός μέλος. Γιατί, διότι οποιοδήποτε ειδικό μπορεί να σας πει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κανονισμού του Δουβλίνου όπως έχει σήμερα είναι ότι αν είναι πολύ καταναγκαστικό δεν φέρνει αποτελέσματα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και με του ετούντε. Προσφέροντα λοιπόν κάποια επιλογή που δεν είναι πλήρω ελεύθερη, αλλά είναι τουλάχιστον κάποια επιλογή μεταξύ των έξι κρατών μελών που δεν μπορούν να προκαθοριστούν, αλλά τη στιγμή τη αίτηση είναι αυτά που έχουν καλύψει το μικρότερο δυνατό βαθμό τη ποσοστώση, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να υπάρχει μια συνοχή, ένα αποτελεσματικό ανθρώπινο σύστημα αντιμετώπιση των περιπτώσεων ασύλου. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, it's, um, Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον, διότι την ώρα που σας άκουγα απέναντι και κάποιες σημειώσεις. Ε, διαπίστωσα ότι κάποια από τα πράγματα που είπατε ε, έρχονται σε αντίθεση με αυτά που είπε η κυρία Μουσολίνη προηγουμένως ε, το θέμα της οικογενειακή επανένωση, παραδείγματο χάρη ίσως στη συνέχεια να σας θέσω κάποιο ερώτημα επ' αυτού διότι από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχει διαφωνία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το εξετάσουμε πρώτα όμως θα δώσω το λόγο στη Λάουρα Φεράρα από τον EFDD παρακαλώ Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη και εγώ για την καθυστέρηση. Έφτασα καθυστερημένο στο αεροδρόμιο. Εδώ και καιρό ζητάμε αναθεώρηση του Δουβλίνου. Εμείς διαφωνούσαμε κάθετα μετά όσα δήλωνε αρχικά ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ε, σε σχέση με το ότι ο κανονισμός του Βλήνου ήταν μια χαρά και ότι πρέπει να περιμένουμε να εφαρμοστεί για να επαληθεύσουμε τι αποτελέσματα είχε εμείς από το 2014 που μπήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσαμε άμεση αναθεώρηση διότι ήταν σαφές ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό της αρμόδιας χώρας για την εξέταση του αιτήματος ασύλου ήταν άνισα, ε, ε, δεν ήταν δίκαια και δεν ε, τηρούσαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 80 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου προβλέπεται συνεργασία και ίση κατανομή των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών μελών. Η μεταρρύθμιση είναι εδώ σήμερα, παρουσιάστηκε πέρυσι αυτό το πακέτο μεταρρύθμισης ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου. Δυστυχώς όμως η μεταρρυθμίση αυτή που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιθυμούσαμε εμείς. Ειδικότερα όσον αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιολιστικής προσέγγισης για τη Μεσόγειο. Ήταν μια έκθεση που προσπαθούσαν να διευκρινίσει από όλε τι απόψει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το τι αναμέναμε απόψη μεταρρύθμιση ε, του ολόκληρου του συστήματο ε, ασύλου τη Ευρώπη. Η μεταρρυθμιστική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να επιτύχει δύο στόχου. Καταπολέμηση τη παράτυπη μετανάστευση και καταπολέμηση των δευτερογενών μετακινήσεων. Κατά την άποψή μου, λείπει κάτι δεν έχουμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο ελέγχουμε τη... γιατί για ποιο λόγο υπάρχουν δευτερογενείς μετακινήσεις και παράτυπη μετανάστευση. Και γιατί αφού διαπιστωθούν τέτοια φαινόμενα υπάρχει κάποια τιμωρητική αντιμετώπιση αλλά δεν έχουμε προσπαθήσει να καταλάβουμε ή δεν έχουμε θελήσει να καταλάβουμε γιατί, ποιες είναι οι αιτίες. Προφανώς ε, η καταπολέμηση της ε, παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί μια νόμιμη εναλλακτική λύση, κάτι που λείπει σήμερα ώστε όποιο προσπαθεί να ξεφύγει, γιατί ξέρετε, όποιο προσπαθεί να ξεφύγει από πόλεμο ή δίωξη, δεν έχει νομικό τρόπο, νόμιμο τρόπο πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να το επιτρέπει να έρθει ασφαλώς στην Ευρώπη. Και ήδη μετά έγραφα στο χέρι του. Όσον αφορά τι δευτερογενεί μετακινήσει, γιατί έχουμε τέτοιε μετακινήσει, διότι προφανώ όπω είπε και η συνάδελφο Σλάιν πριν από μένα, πρόκειται για ανθρώπου, πρόκειται για ετούντε άσυλο που γνωρίζουν καλά τον κανονισμό του Δουβλίνου και ξέρουν ότι αν υπάρχουν συγγενεί αλλού, αν θέλουν να πάνε σε αυτού, σε ένα άλλο κράτο μέλο, υποχρεούνται παρόλα αυτά να παραμείνουν ένα-δύο χρόνια στην πρώτη χώρα άφηξη παρότι δεν ήταν ε, ο προορισμός τους αυτή η χώρα. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους ετούντες άσυλο, αλλά και στις πρώτες χώρες άφηξης. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ιταλία, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε διαπιστώσει πώς λειτουργήσε, μάλλον δεν λειτουργήσε ο, ο μηχανισμός υποστήριξης Ελλάδας και Ιταλίας με τη μετεγκατάσταση που θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες με ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά αρνητικό. Ε, λιγότεροι από 5.000 ε, ετούντες άσυλο έχουν μετακατασταθεί από την Ιταλία και ε, λίγο παραπάνω από τους 12.000 έχουν μετακατασταθεί από την Ελλάδα όταν 160.000 ήταν οι ετούντες άσυλο και κατάσταση. Είναι γελία λοιπόν τα ποσοστά αυτά και απεικονίζουν τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόταση μεταρρύθμισης του Δουβλίνου. Εμείς εκεί έχουμε υποβάλει σχεδόν 170 τροπολογίες, δηλαδή ξαναγράψαμε ουσιαστικά τον κανονισμό. Με σκοπό να αναδείξουμε τα σημαντικά σημεία, αυτά που ονομάζουμε κόκκινε γραμμές. Πρώτα απ' όλα το θέμα του κριτηρίου της πρώτης χώρας ε, άφηξης ε, εισόδου ως ε, χώρας αρμόδιας για την διεκπαιρέωση της αίτησης ασύλου. Αυτό αυτή η αρχή πρέπει να εξαφανιστεί γιατί αυτή οδήγησε στι τεράστιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ιταλία και η Ελλάδα και είναι και η αιτία των δευτερογενών μετακινήσεων. Ο μηχανισμό ε, κατανομή των ετούντων άσυλο δεν μπορεί να είναι φιλανθρωπικό μηχανισμό ούτε μηχανισμό αλληλεγγύη που να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκης ε, βάσει εκτιμήσεων τη Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Είναι μια κατάσταση που δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες, ακόμα περισσότερες από ή αυτές που ήδη αντιμετωπίζουν Ιταλία και Ελλάδα για μα. ο μηχανισμό καταμερισμού των ετούντων ασύλο πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα και να είναι υποχρεωτικό. Οι τροπολογίε λοιπόν που έχουμε υποβάλει κινούνται προ αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατάργηση, η κατάργηση τη ε, χώρας πρώτης εισόδου και η αυτόματη ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης κατανομής. Πώ θα ενεργοποιείται βάσει των τροπολογιών που έχουμε υποβάλει θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή επανένωση αυτό διότι εγώ προσωπικά έχοντας ε, ταξιδέψει σε όλη την Ιταλία και σε άλλα κράτη-μέλη έχω πάει στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Σουηδία, στην Ελλάδα και διαρκώς μας καταγγέλουν ότι όσοι θέλουν να επανενωθούν με τους συγγενείς τους συγγενείς τους που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη ε, ξαφνικά μπλοκάρονται στην Ιταλία ή στην Ιταλία, στην Ιταλία στην Ελλάδα συγγνώμη, για χρόνια ή για μήνες. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. Εμείς λοιπόν με τις τροπολογίες μας θέτουμε αυτό ως πρώτο κριτήριο προς εφαρμογή. Με διεύρυνση μάλιστα της έννοιας της οικογένειας σε σχέση με την αρχική έννοια. Γιατί, διότι έτσι εξασφαλίζουμε επανένωση, μεγαλύτερη ένταξη καλύτερο καταμερισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους ετούντε άσυλο. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς σε άλλα κράτη-μέλη, εκεί ενεργοποιείται ο μηχανι... αυτόματος ο αυτόματος και υποχρεωτικός μηχανισμός που βασίζεται σε ποσοστώσεις, ποσοστώσεις που βασίζονται σε πληθυσμό, σε καθάριστο εγχώριο προϊόν ε, και αυτά είναι τα τρία κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι ποσοστώσεις των ετούντων άσυλο που κάθε κράτο θα πρέπει να υποδεχθεί και θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο βάσει των αλλαγών πληθυσμού, ανεργία και ΑΕΠ. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Τώρα, ε, επειδή σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο μηχανισμός προτείνουμε κυρώσεις. Δηλαδή διακοπή των διαρθρωτικών ταμείων ή των ταμείων συνοχής. Γιατί? διότι η πρόταση της Κομισιόν ε, ε, αποσκοπούσε σε ε, τιμωρία του κράτους μέλους με 250.000 ευρώ για κάθε ετούντα άσυλο που δεν έχει γίνει δεκτός. Για εμάς το μέτρο αυτό δεν είναι σωστό. Πρώτον, μας φαίνεται ότι ποσοτικοποιεί οικονομικά την αξία ενός ανθρώπινου όντως ηθικά θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό. Και δεύτερον, διότι πολύ δυστυχώς ε, κάποιες κυβερνήσεις μπορεί να αποφασίσουν να πληρώσουν εις βάρος των πολιτών τους, να πληρώσουν το πρόστιμο αυτό και να μην ε, ε, εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Όταν κόβονται διαρθρωτικά ταμεία που έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλά κράτη-μέλη για αναγέννηση της οικονομίας τους. Ε, εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει από καλό αποτρεπτικό μηχανισμό. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες του ετούντος, ε, οι γλωσσικές γνώσεις, η ύπαρξη κάποιων σχέσεων ε, με νόσεις, με οργανώσεις όπου θα μπορούσε να ενταχθεί καλύτερα για να καθοριστεί ποιο κράτος μέλος θα μπορούσε να είναι αρμόδιο. Ε, βάσει φυσικά πάντα των ποσοστώσεων. Αυτά είναι τα κύρια σημεία τα οποία εμείς προβλέπουμε με τις δικές μας ε, τροπολογίες ε, και οι γραμμές που θα ακολουθήσουμε εμείς για τη θέση μας όσον αφορά τον κονισμό του Δουβλίνου. Εμείς δεν ζητάμε φιλανθρωπική αλληλεγγύη, επαναλαμβάνω. Ζητάμε να τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει μια διασφάλιση της συνεργασίας, να αντιμετωπιστεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ευρωπαϊκό τρόπο και όχι αφήνοντα την ευθύνη μόνο σε μερικα Εύχομαι λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε κάποια συνένεση και κάποια υποστήριξη πρώτον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεύτερον κυρίως από το Συμβούλιο στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον που αναφέρατε την παρακράτηση διευθυντικών ταμείων αντί για πρόστιμο. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα την οποία ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Βίκστρομ. Θα δώσω το λόγο ε, για να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Θα ακούσουμε τρεις και κατόπιν ε, τις απαντήσεις και μετά άλλες τρεις κλπ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο πρώτα εσείς. Παρακαλώ. Έχω νέα ερώτηση τώρα που άκουσα τις δύο κυρίες από την Ιταλία. Το όνομά σας παρακαλώ και από πού, έρχεστε. Μαρή Από ε, την ε, γερμανική τηλεόραση ARD. Οι κυρίες από την Ιταλία ε, τόνισαν το θέμα της ευθύνης και αναφέρθηκαν και στο σύστημα καταχώρησης. Για την ε, Ιταλία και ιδιαίτερα για την Ελλάδα αυτό είναι θέμα κλειδί, η καταχώρηση. Κυρία Σλάιν, είπατε ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται στην πρώτη χώρα άφηξης ε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Ιταλία η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί ακριβώς να πετύχει αυτό. Τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν όσον αφορά το σύστημα καταχώρησης. Δεν λειτουργεί όμως. Τι ιδέες, τι προτάσεις έχετε για να γίνει πιο λειτουργικό το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κοτσίνσκι, από την Πολωνία. Μία ερώτηση προς την κυρία Βίκστρομ και την κυρία Φεράρα σχετικά με την ε, παρακράτηση των διαρθρωτικών ταμείων. Η Πολωνία, η Αυστρία και η Ουγγαρία η Πολωνία όχι τόσο πολύ, αλλά η ε, Αυστρία και η Ουγγαρία κλονίστηκαν από άφηξη χιλιάδων ε, μεταναστών και είχαμε ε, τεράστιες ε, πολιτικές ε, αναταραχές στην Αυστρία κατέρευσε η κυβέρνηση λόγω της κρίσης αυτής και γι' αυτό η χώρα αυτή δεν θέλει να υποδεχθεί μετανάστες διότι φοβάται ακριβώς τι θα γίνει. Η Αυστρία και η Ουγγαρία λοιπόν που ήταν οι πρώτες χώρες που άρχισαν ε, να λένε ότι θα πρέπει να αρνηθούμε την είσοδο σε ανθρώπους ε, που ε, πάνε προς την Γερμανία. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να τιμωρήσετε την Αυστρία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολύ σωστή ερώτησή σας. Παρακαλώ. Αλφόνσο Μπιάνκη από την Ιταλία. Κάνω clarification, because Mrs. Mussolini talked about... Καταρχάς, σε μια διευκρίνηση, η κυρία Μουσολίνη ανέφερε ότι η συμπερίληψη του θέματος ε, της αλλαγής του κλίματος ε, στο θέμα περί ασύλου αυτό είναι πρόταση της κυρίας Βίκστρομ ή βρίσκεται στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης θα ήθελα να ακούσω από τους ευρωβουλευτές που είναι ακόμα εδώ πώς βλέπουν το θέμα της παροχής ασύλου σε ανθρώπους ε, που μετακινούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω των απειλών της ε, κλιματικής αλλαγής. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Ναι, το θέμα της κλιματικής αλλαγής αυτό δεν συνδέεται με την πρόταση του Δουβλίνου. Αυτό έχει να κάνει με, τις, την τροποποίηση στην οδηγία για τις δεξιότητες οι οποίες θέλουν να γίνουν κανονισμός. Ε, δηλαδή δεν σχετίζεται άμεσα με το Δουβλίνο. Τώρα, είναι αλήθεια ότι το ΕΛΚ δυσκολεύεται με αυτό και δεν είναι η μόνη διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει όμως ε, ένας συμφωνημένος διεθνής ορισμός, ένα συγκεκριμένο καθεστώς για τους κλιματικούς ε, πρόσφυγες ή ε, ε, ψάχνουμε έναν ορισμό που να γνωρίζει το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν έχουμε ακόμα, δεν το έχουμε ακόμα καταφέρει. Και η Τάνια Φάγεν από το S&D είναι η συγκίτρια για το σχετικό κείμενο μια και έχω το μικρόφωνο, να πω κάτι για τα διευθυντικά ταμεία. Δεν υπάρχει συμφωνία από αυτού. Είναι ένα θέμα προσυζήτηση. συζήτηση. Όμως, ε, επί της αρχής, ε, αυτό που ισχύει είναι η αλληλεγγύη, η αρχή της αλληλεγγύη που υπάρχει στη συνθήκη. Νομίζω όλοι το είπαν, όλες οι πολιτικές ομάδες. Το θέμα είναι πώς θα συνεργαστούν τα κράτη-μέλη από αυτού. Υπάρχει το θέμα τη διαφοράς μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας, που χάρη το 2015, που εφάρμοσαν άλλο κομμάτι της, του, του Δουβλίνου. Υπάρχει μια ρήτρα ε, κυριαρχίας που μπορεί μια χώρα να πει εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα άτομα που είναι στο έδαφος μας. Και γιατί την, κατ' εμέ αυτό είπε η Γερμανία. Ε, και κάποιοι αυτό το κατεξέλαβαν ω πρόσκληση. Η Ουγγαρία εφάρμοσε ε, τον κανόνα τη πρώτη χώρα εισόδου Γι' αυτό είχαμε και την ένταση. Ε, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ξαφνικά ε, να υψώσουν τύχη αντί να κάψουν γύρω από ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν γύρω από ένα μηχανισμό αλληλεγγύης. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχουμε να κάνουν με τη διαφορά ερμηνείας. Ε, αυτό που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε είναι να κρατήσει σαφέ ότι το να μοιραστούμε τις ευθύνες είναι αυτό που μετράει. Πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αυτά τα οποία συμφώνησαν στο άρθρο 18. Ναι, η Γερμανία όμως καλούσε τους ε, ε, μετανάστες ε, στην Ευρώπη λέει ο δημοσιογράφος. Ακούστε, λέει η κυρία Λάμπερτ, εγώ αυτό που κατάλαβα από το που είπε η κυρία Μέρκελ είναι ότι δεν, πρόκειται, δεν πρόκειται να επιστρέψει, να στείλει πίσω ανθρώπους. Και αυτό ε, το είδαν οι άνθρωποι αυτοί ως μια ευκαιρία. Ε, είναι από τις λίγες φορές ε, στην ζωή μου που έχω κατέβει στους δρόμους στο Λονδίνο σε μια διαδήλωση και έχω δει ανθρώπους ε, που να ε, συγχαίρουν τη Γερμανία για κάτι που έχει κάνει γιατί να τους κατηγορούν που κέρδισαν πάλι το παγκόσμιο κύπελο. Ε, εν περιπτώσει, είναι πολύ θετικό που η Γερμανία είπε σε άλλες χώρες, εδώ υπάρχει ζήτημα, πρέπει να βοηθήσουμε. Ε, τώρα βεβαίω πολλές άλλες χώρες δεν ακολούθησαν αυτήν την όδο και ύψωσαν τα τείχη που ελπίζαμε το 1989 είχαν εκλείψει. Μάλιστα. Κάποιος άλλος. Έγινε ένα ερώτημα από μια Γερμανή δημοσιογράφο, νομίζω προς εμένα, για το σύστημα καταγραφής. Ακούστε, αυτή τη στιγμή υπάρχει την προσέγγιση με τα hot spot στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Ήμουν στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα μια αποστολή με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και νομίζω επισκεφτήκαμε όλα τα hot spot σχεδόν δεν έχω πιστεί και τόσο από την προσέγγιση. Στην Ιταλία δεν υπάρχει επαρκή νομική βάση. Ε, χρειάζεται νόμος για να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο. Δεν αρκούν δηλαδή οι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια μέρη όπου οι άνθρωποι είναι περιορισμένοι. Έτσι. Είναι, στη Λαπεντούς είναι κλειστό ε, το κέντρο αυτό. Ε, τώρα από εκεί πέρα το γεγονός ότι υπάρχει παρουσία ευρωπαϊκών φορέων στα hotspot που βοηθούν κατά την καταγραφή, η ΕΑΣΟ, Frontex, ε, που βοηθούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, ε, τα τελικά αποτυπώματα των ε, μεταναστών που φτάνουν. Δεν, βλέπω, δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι αυτό δεν λειτουργεί. Σε πέδο εγγραφή, σε πέδο καταγραφή, το ποσοστό καταγραφή έχει ξεπεράσει το 90%. Έτσι, ό,τι φορά λοιπόν την αποφυγή αυτού που συνέβαινε νωρίτερα, ότι πολλοί δηλαδή ετούντες ε, δεν ε, καταγραφόταν ε, και τελικά πήγαιναν σε άλλες χώρες, ε, Τώρα το ποσοστό είχε αυξηθεί το ποσοστό εγγραφή. Τώρα προσπαθούμε να έχουμε ένα πιο καλό, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα, εφόσον αυτό ρωτάτε. Ε, προσπάθησα να το πω και προηγουμένω. Μπορεί να φαίνεται προκλητικό, αλλά δεν είναι. Ο καλύτερο τρόπο για να αποφύγουμε τι δευτερογενεί μετακινήσει, το είπε και η Λάουρα, είναι να πάψει να ισχύει το κριτήριο της χώρας, της πρώτης χώρας εισόδου. Γι' αυτό το λόγο κάποιες χώρες δεν είναι και τόσο ακριβείς κατά την εγγραφή και την καταγραφή των μεταναστών στο παρελθόν. Και αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι ετούντες αρνούνται, αρνούνται να καταγραφούν. Γνωρίζουν το, τι, λέει, το Δουβλίνο, δεν έχουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα κάποιον συγγενή και ξέρουν ότι αν ε, καταγραφούν στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ε, την περσμένη εβδομάδα ε, είδαμε 15χρονα κορίτσια τα οποία φύγαν μόνα τους από το Χαλέπι και βρίσκονται σε ένα νησί και περιμένουν να ξαναδούν τη μητέρα τους με το σύστημα ε, επανένωση. Με ένα τέτοιο σύστημα εγώ δεν τους κατηγορώ. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Εμείς λοιπόν οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί. Τι λέμε λοιπόν. Αυτό το κριτήριο λοιπόν της πρώτης του πρέπει να εκλείψει, να έχουμε ένα κεντρικό ενιαίο σύστημα. Μιλάμε για ανθρώπου που έχουν δικαιώματα, έχουν δικαίωμα ε, να ζητήσουν άσυλο. Έχουν κάποιες Κάποιου δεσμού με κάποιε χώρες. Μπορεί να έχουν μείνει στο παρελθόν σε μια χώρα, μπορεί να έχουν ένα δίπλωμα από μια χώρα, ε, τη γλώσσα, να γνωρίζουν τη γλώσσα. Να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Και έτσι δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη κάποιο να αποφύγει την πρώτη καταγραφή και να περνάει στη δευτερογενή μετακίνηση. Μπορεί κάποιο να μην φτάσει τελικά στο, στη χώρα στην οποία ενεργόταν να πάει, αλλά είναι ένα σύστημα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν, μπορούν να πούν πού είναι η οικογένειά του, ε, πού έχουν δεσμού και εντό ενό μήνα, εφόσον δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο κριτήριο για αυτού, τότε μπαίνουν στο το, μηχάνισμα, το, το μηχανισμό συγγνώμη, δίκαιης κατανομής. Ε, από την εμπειρία μου στη Λαμπεντούσα, όπου μιλούσαμε με του ανθρώπου αυτού που έφταναν, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει λόγος από εκεί και πέρα κάποιος να εξαφανιστεί και να προβεί σε μια δευτερογενή μετακίνηση. Ε, και κάτι ακόμα. Κάτι, έγινε μια ερώτηση για τους κλιματικούς πρόσφυγες. Θα πρέπει, είναι καιρό σε διεθνές επίπεδο να το, το δούμε αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τους κλιματικούς πρόσφυγες. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Βεβαίως ε, στο μέτρο του δυνατού πρέπει να κάνουμε το ίδιο και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά είναι κάτι που, όπω είπε και η Τζιν, ε, εξετάζεται στο φάκελο για τα qualifications και όχι στη συζήτηση για το Δουβλίνο. Και το ρεύμα τη Πολωνία να προσθέσω κάτι. Ακόμα συζητούμε το θέμα των ενδεχόμενων κυρώσεων προ τα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν και δεν ε, τι δεσμεύσει. δεσμεύσεις Να πω όμω κάτι. Η βασική αρχή είναι η εξή. Δεν μπορείτε να έχετε μόνο τα ωφέλη του να συμμετέχετε σε μια μεγάλη ένωση και ποτέ να μην μοιράζεστε τις ευθύνες. Αυτό το κάνουν παιδάκια, ε, πεντάχρονα. Δεν το κάνουν κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών. Τα διορθωτικά ταμεία είναι άλλη, ένα πρόσωπο της αλληλεγγύης, αλλά όταν μιλάμε για την μετάσταση και το άσυλο, είδαμε στην Ιταλία και στην Ελλάδα ότι η οικονομική συνεισφορά δεν αρκεί. Πρέπει κάποιο να αναλάβει την ευθύνη και, και σε ό,τι φορά την εξέταση του ζητήματο. Δεν μπορούμε αυτέ τι χώρε να καταλήψουμε και να γίνουν ε, τεράστια στρατόπεδα προσφύγων επειδή κάποιες χώρες ε, διστάζουν να κάνουν το μέρος της δουλειάς που τους αναλογεί. Να μην ξεχνάμε ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν δίνει ε, αυτόματα το καθεστώς πρόσφυγα σε κάποιον. Λέει όμως σε ποιο κράτος μέλος, ποιο κράτος μέλος αναλογεί η ευθύνη να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Από εκεί και πέρα, σε διεθνές επίπεδο πρέπει να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί καθεστώς ασύλου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να μιλήσω ιταλικό, ιταλικά για μία φράση μόνο. Say in Italian is that... Στα ιταλικά λέμε δεν υπάρχει μία αιτία στον κόσμο δεν έχει γραφτεί πουθενά ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δεν έχει γραφτεί πουθενά και ότι πρέπει να επιφορτιστούν με τι αιτήσει ασύλου, που είναι πολυάριθμε, που σημαίνει διοικητικό φόρτο, γραφειοκρατικό φόρτο, οικονομικό φόρτο, που οδήγησε σε κατάρρευση το σύστημα υποδοχή ορισμένων κρατών. Πουθενά λοιπόν δεν είναι γραμμένο ότι μόνο δύο, τρει, τέσσερι χώρε, κράτη-μέλη, πρέπει να υπομισθούν όλη τη δουλειά για λογαριασμό όλων. Ευχαριστώ λοιπόν εν συντομία για να απαντήσω στις τρεις ερωτήσεις ε, που τέθηκαν όσον αφορά τη Γερμανίδα δημοσιογράφο που ρώτησε για την ευθύνη καταγραφής γιατί δεν λειτουργεί και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις γιατί δεν λειτουργεί πρώτα απ' όλα πολύ πρακτικά δείτε το τη στιγμή που κάποιος φτάνει με ε, ένα σκάφος στην Ιταλία ε, έχουν δημιουργηθεί αυτά τα hot spot. Έχουμε έξι hot spot, σύνη, Μινέο, Λαμπεντούζα, Τράπανη, Τάραντο, αλλά ο κόσμο δεν φτάνει μόνο εκεί που υπάρχουν τα hot spot αυτά. Τα 6-7 hot spot φτάνουν και στην Καλαβρία, στην Καμπανία, ε, στη Σαρδινία, όπου δεν υπάρχουν hot spot. Στο χρονικό πλαίσιο λοιπόν μεταξύ της ε, άφηξης ε, στην ακτή και της άφηξης στο hot spot χάνεται πολλοί κόσμος. Οπότε πρακτικά η πραγματικότητα είναι τέτοια που πολλοί κόσμος δεν καταγράφεται. Ο κόσμος ε, χάνεται, εξαφανίζεται. Γιατί, γιατί ξέρει ότι με το που καταγραφεί στην Ιταλία υποχρεούται να παραμείνει εκεί. Αυτά είπαμε και πριν. Παρόλε τι προσπάθειε λοιπόν τη Ιταλία και την καλή θέληση και τη δημιουργία των hot spot, παρόλα αυτά η κατάσταση παραμένει διότι η βάση η νομοθετική του κανονισμού του Δουβλίνου είναι λανθασμένη. Αν δεν τη λύσουμε λοιπόν, αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν ετούντες άσυλο που, τους, ε, που χρειάστηκε να τους αναγκάσουμε να τους πάρουμε τα τελικά αποτυπώματα ε, ή μάλλον που ε, έσπασαν τα χέρια τους για να μην δώσουν ε, δακτυλικά αποτυπώματα. Άλλοι που αρνήθηκαν καταγραφή. Ε, φτάσαμε σε στιγμές που αναγκαστήκαμε να αναγκάσουμε ανθρώπους να, τους, να, βάλουμε τα χέρια τους πάνω στα μηχανήματα για να πάρουμε τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Λειτουργεί λοιπόν αυτό το δουβλίνο, ε, το σύστημα των hotspot ή όχι, όταν αναγκάζουμε ανθρώπους έτσι. Υπάρχει πέραν της θεωρίας και μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να γνωρίζουμε από πρακτική άποψη. Και βάσει αυτών μετά πρέπει να ψηφίζουμε. Ποιε είναι οι λύσει. Η λύση είναι να αλλάξουμε το Δουβλίνο, να μην υποχρεώνουμε του ανθρώπου που φτάνουν στην Ιταλία στην Ελλάδα να παραμένουν στην Ιταλία στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα είναι πιο διατεθειμένοι να καταγραφούν γιατί θα ξέρουν ότι δεν υποχρεώνονται να παραμένουν εκεί θα ξέρουν ότι μπορούν να πάνε σε άλλα κράτη-μέρη. Και αυτό θα διευκολύνει και την Ιταλία που παρά τις βοήθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΑΣΟ, τη Frontex, την Ευρωπόλ, παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να τα κάνει όλα μόνη τη. Για να απαντήσω στην ερώτηση περί παρακράτησης των διαρθρωτικών ε, ταμείων, ε, δεν πρόκειται για κάποια τροπολογία ε, τιμωρητική προς την Αυστρία, την Ουγγαρία, που οι κακομοίρε το 2015 έλαβαν τόσους πολλούς διερχόμενους ε, τον Τεσάσιλο και δεν τους θέλουν πια γιατί αυτό το εγωιστικό λόγο θα μπορούσε να έχει και η Ελλάδα, η Ιταλία. Έφτασαν τόσοι πολλοί από το 2015 και το 2016 που δεν τους θέλουμε πια. Εμένα μου φαίνεται ότι το να λέτε τέτοια πράγματα είναι ε, ε, αβάσιμα ουσιαστικά. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα όταν μιλάμε για μια κοινότητα, για μια ένωση, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι αντιμετώπισαν δυσκολίες. Η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, οι 7-8 χώρες από τις 27 πλέον που έλαβαν, ε, ανέλαβαν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και η διαχείριση αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη το 2015 και το 2016, όπου μεγιστοποιήθηκαν οι ροές. Η τροπολογία αυτή λοιπόν δεν αποσκοπεί να πλήξει την Αυστρία ή την Ουγγαρία, αλλά να τιμωρήσει τις χώρες που δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τις χώρες που από τη μια πλευρά παίρνουν χρήματα, αλλά από την άλλη δεν θέλουν να δώσουν τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τον τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Τρία-τέσσερα λεπτά μας μένουν για αυτό το τμήμα της συζήτησης. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο. Νεγκουίντο Ρότολο, Ιταλία από την Τίσκαλη. Στις 3 Οκτωβρίου του 2013 έχουν περάσει τέσσερα χρόνια στις παραλίες της Λαμπεντούζα περισυλλέχθησαν 366 σώματα χωρίς δάχτυλα και χωρίς ζωή άψυχα και τέσσερα χρόνια μετά η Ιταλία δεν έπαψε να εργάζεται χωρίς καμία αλληλεγγύη από την Ευρώπη για να υποδεχθεί τους ανθρώπους που ερχόνταν από όλα τα μέρη του κόσμου. Ενώ η Ευρώπη λοιπόν και ορισμένες χώρες αποφάσιζαν να αποσταθεροποιήσουν πολιτικές, γεωγραφικές, εδαφικές περιοχές όπως το Ιράκ μετά τη Συρία υποστήριξαν την ε, Αραβική Άνοιξη, συνέβαλαν ε, για την κατάρρευση του Καντάφη, ασχολήθηκαν μόνο με αυτό, αλλά ουδέποτε κατάφεραν να διαχειριστούν ε, όλα αυτά τα αποτελέσματα, διότι όλοι οι άνθρωποι που έφτασαν έτσι για αυτούς τους λόγους στην Ευρώπη έφτασαν για ένα λόγο, για πολιτικό λόγο και η Ευρώπη προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση αλλά ε, και βάσει των όσων ακούσαμε μέχρι στιγμής αντιλαμβάνομαι ε, ανικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει το θέμα. Εγώ ως Ιταλός έχω να πω ότι εμείς ασχοληθήκαμε με τους μετανάστες στις 3 Οκτωβρίου, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια ε, Τώρα έχουμε τις ΜΚΟ που πηγαίνουν στα εγχώρια έδατα της Λιβύης για να πάρουν τους ανθρώπους που φεύγουν από τη Λιβύη, τους μετανάστες. Και εκεί συμμετέχουν πολύ πολλές ευρωπαϊκές εθνικότητες. Γιατί τους φέρνουν πάντα στην Ιταλία, γιατί δεν τους πάνε στη Βαρκελόνη, γιατί τους πάνε αλλού. Και έρχονται πάντα στην Ιταλία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί είσαστε τόσο βέβαιοι ότι έχει αποτύχει το σύστημα του ε, Δουβλίνου, διότι πριν δύο χρόνια δεν ε, ε, θεωρεί το αποτυχημένο. Απέτυχε επειδή κάποια κράτη-μέλη δεν πληρούσαν τις υποχρεώσεις τους ή επειδή άνοιξαν όλες τις πόρτες, δηλαδή και πάλι δεν πληρούσαν τις υποχρεώσεις τους. Γιατί λοιπόν θεωρείτε ότι απέτυχε το σύστημα και όχι κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες. Και επίσης, γιατί ε, εφόσον έχετε ε, δεχτεί την προσχώρηση Δέκα επιπλέον ε, κρατών μελών. Ε, έχετε πρόσβαση στις ε, αγορές τους, στις οικονομίες τους. Γιατί τώρα πια θεωρείτε ότι δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ακόμα ερώτηση και κατόπιν θα κλείσουμε. question. Μία ερώτηση έχω. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 60.000 πρόσφυγες που δεν θέλουν να παραμείνουν στη χώρα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πότε θα μετατρέψετε τη θεωρία σε πράξη. Πότε θα τους δώσετε τη δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο, να μεταφερθούν κάπου αλλού. Διότι αυτή τη στιγμή απλά περιμένουν. Thank you very much. Um, I would ask you to take... Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη, σίγουρα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις διότι η απάντηση θα πρέπει να δοθεί με ευρωπαϊκούς όρους και όχι εθνικού, όπως είχε γίνει μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή η απάντηση υπήρξε εθνική. Τώρα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Θα τα καταφέρουμε ή όχι. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δύο χρόνια. Μέχρι στιγμή δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει. Μέχρι στιγμή υπάρχουν τόσα πολλά κενά ξεκινώντας από την έλλειψη νόμιμων οδών πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για καταπολέμηση της παράτυπη μετανάστευσης, καταπολέμηση των διακινητών ε, ανθρώπων. Μα τι απλούστερο από το να προσφέρουμε μία νόμιμη εναλλακτική σε όποιον ξεφεύγει από πολέμους, διαφεύγει από πολέμους και διώξεις. Όταν οι άλλοι τους, η μόνη λύση που έχουν είναι να πληρώσουν εμπόρους, διακινητές, ε, ε, για να βρεθούν ε, σε σώο έδαφος ε, περνώντας τη Μεσόγειο με ένα φουσκωτό ή με, περνώντας μέσα από ένα φορτηγό ψυγείο όπως έγινε τις προάλλες με κάποιους ανθρώπους που πέθαναν μέσα ένα φορτηγό ψυγείο είναι παράδοξο να λέμε ότι κάποιος ταξιδεύει και πληρώνει για να ταξιδέψει υπό τέτοιες συνθήκες για να σωθεί αυτό είναι το παράδοξο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Υπάρχουν ελλείψει κενά ε, νομικά τέτοιου τύπου και αφορούν ε, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν αφηθεί πλέον στη ΜΚΟ. Έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση Μαρενόστρουμ. Μετά από αυτήν την επιχείρηση που ήταν Ιταλική επιχείρηση με κόστος που η Ιταλία δεν μπορούσε πια να υποστηρίξει μόνη της. Αυτή η επιχείρηση δεν αντικαταστάθηκε από αντίστοιχη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Οπότε τηρούμε τους κανόνες της θάλασσας. Παρέχεται ε, διάσωση τη στιγμή που ε, εκπέμψει, ε, ακούστε ένα SOS, πάμε να σώσουμε ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχουν στοχευμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνες και διάσωσης. Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάχιστα. Και μάλιστα θα έπρεπε να επιταχύνει λίγο, διότι αλλιώς θα μείνουμε στην ιστορία ως ε, ικανοί μόνο να σηκώνομαστε όρθιοι και να, κάνουμε, να τηρούμε ένας υγιή και τίποτα άλλο. Γιατί μιλάμε για αποτυχία του Δουβλίνου και όχι για τις ευθύνε των κρατών μελών. Ε, έτσι συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Πρέπει να μιλάμε ε, ως Ευρώπη. Πρέπει να λέμε τι πρέπει να κάνουν όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο 7-8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αποτελείται από 27 κράτη-μέλη. Μέχρι σήμερα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ε, έχει αφαιθεί στα χέρια 7-8 χωρών. Οι υπόλοιπε 20 δεν έχουν συμβάλει καθόλου και με κανένα τρόπο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Δεν λειτουργεί δηλαδή ο κανονισμός του Δουβλίνου διότι αυτός ο κανονισμός αποθέτει στα χέρια ελάχιστον κρατών μελών την ευθύνη των μεταναστευτικών ροών. Οι υπόλοιπε 20 χώρε που σήκωσαν τα χέρια ψηλά το έκαναν νόμιμα, διότι αυτό προέβλεπε το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο προέβλεπε ότι η πρώτη χώρα εισόδου είχε την ευθύνη να διεκπαιρεώσει τις αιτήσεις ασύλου. Οπότε έλεγαν εγώ δεν ε, έχω να κάνω τίποτα, είμαι απελαγμένος, δεν έχω καμία ευθύνη. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε την προσοχή μας στον κανονισμό του Δουβλίνου, γιατί αυτός ε, είναι ε, η νομική βάση, βάση της οποίας όλων των, όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν ε, ίσες ευθύνες. Και έτσι δημιουργείται η ανισορροπία αυτή που παρατηρούμε όσον αφορά τις ευθύνες. Okay, ehm, Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην ερώτηση του πρακτορείου Τίσκαλη. Λοιπόν, τι έχει κάνει η Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει διατυπωθεί σωστά η ερώτηση. Γιατί πρέπει να δούμε τα πράγματα όπω έχουν. Εδώ και 20 χρόνια μιλάμε για κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που έχουμε καταφέρει να θέσουμε ε, σε, κοινό, σε κοινή χρήση είναι ένα τεράστιο νεκροταφείο στη Μεσόγειο που είναι ευρωπαϊκή θάλασσα, δεν είναι ιταλική ούτε ελληνική. Μόνο αυτό καταφέραμε να υλοποιήσουμε. Α δούμε τα στοιχεία που είπε και η Λάουρα. Μόνο 7-8 κράτη-μέλη τόσα χρόνια αντιμετώπισαν μόνα του το 80% των αιτήσεων ασύλου σε ολόκληρη την Ένωση. Αντιλαμβάνεται κανεί λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι τι έκανε η Ευρώπη, ούτε πού είναι η Ευρώπη μπροστά σε όλες αυτές τις τραγωδίες ε, ε, που εκτελήσονται στις ακτές της Σικελίας αλλά όχι μόνο, όχι μόνο και στις ακτές της ε, Πούλια και της Καλαβρίας. Το θέμα είναι πού είναι οι άλλες 20 κυβερνήσεις. Τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Οι άλλες 22 κυβερνήσεις. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, διότι ξέρετε, το Σαββατοκύριακο πάμε όλοι σπίτι μας Έχω την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα επίπεδα ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σαφέ λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο από τον Απρίλιο του 2015, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το παρόν Κοινοβούλιο, ζητά ε, σύστημα αυτόματο και μόνιμο μετεγκατάσταση. Απαιτεί κάθε κράτο μέλο να συμμετέχει στο βαθμό που του αναλογεί. Ζητά, για παράδειγμα, νόμιμες ασφαλείς οδού πρόσβαση. Ζητά η Ελλάδα και η Ιταλία να μην αφαιθούν μόνε του. Άλλο θέμα τώρα είναι ο εθνικός εγωισμός που παρατηρούμε στις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Άλλο θέμα είναι η Επιτροπή που μετά από την τραγωδία αυτή που υπενθυμίσατε εσείς αλλά και τις άλλες που ακολούθησαν τον Απρίλιο του 2015 με 950 νεκρούς δεν θυμάστε εκεί η Κομισιόν πρότεινε ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση και μετά το σύστημα μεταγκαταστάσεων. Η Κομισιόν λοιπόν προσπάθησε να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη να συμμετέχουν και να λάβουν τις ευθύνες τους. Και τι πέτυχε μετά από 1,5 χρόνο από τις 160.000 μεταγκαταστάσεις που υποσχέθηκαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υλοποιήθηκαν 17.903. Αυτό ενώ ο Καναδά σε τέσσερις μήνες πέρυσι επανεγκατέστησε στην επικράτειά του 35.000 ανθρώπους με έναν ωκεανό στη μέση. Τι σημαίνει αυτό ότι 27-28 Ευρωπαίοι εταίροι κατάφεραν να επιτύχουν το λιγότερο από το μισό αυτό που κατάφερε να επιτύχει ο Καναδάς. Για να καταλάβετε γιατί νούμερα μιλάμε, γιατί δεν μιλάμε για καμία εισβολή. Έρχομαι και στη δεύτερη ερώτηση, δεν μιλάμε για εισβολή. Το 2015 1.300.000 αιτήσει ασύλου υποβλήθηκαν σε ολόκληρη την Ένωση και αυτή ήταν η χρονιά με τις περισσότερες αιτήσει. Είναι ο αριθμός ε, μεταναστών που έχει υποδεχθεί ο Λίβανος με 3 εκατομμύρια κατοίκους. Μιλάμε για, το 5%, για, το, για ένα τεράστιο ποσοστό της, ε, ε, του πληθυσμού του και στην Ευρώπη μιλάμε για το 0,2%. Κάποιος αναφέρθηκε στη Μέρκελ προηγουμένως και είπε τι έχει κάνει η Γερμανία να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι υποστηρίκτρια της Μέρκελ. Είμαι αντίθετη πολιτικά. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι αν εκείνη τη στιγμή οι άλλες κυβερνήσεις δεν την είχαν αφήσει μόνη της να λέει διασάφεντας θα τα καταφέρουμε, σήμερα δεν θα είχαμε αυξανόμενη ξενοφοβία, ε, δεν θα είχαμε την επιτυχία των ακροδεξιών κομμάτων, διότι η ανικανότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν με κοινέ λύσει αυτή την κοινή πρόκληση δημιούργησε την εντύπωση ότι ήταν μη διαχειρίσιμη. Ότι βρισκόμαστε ενώπιον μια εισβολή, ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη αυτών των Ευρωπαίων ηγετών. Και για να κλείσω, για την Ελλάδα. Α μη συγχαίρουμε τα επίπεδα ευθύνη. Εμεί είμαστε Ευρωπαίοι βουλευτέ, Ευρωβουλευτέ. Έχουμε ψηφίσει πριν από τρει εβδομάδε στο Στρασβούργο καταδικάζοντα τι κυβερνήσει που δεν πραγματοποίησαν τις μετακατάστασεις που υποσχέθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία ζητώντας να κάνουν επιτέλους τη δουλειά τους το πρόγραμμα μετακαταστάσεων από την Ιταλία και την Ελλάδα να παραταθεί ε, μετά από το Σεπτέμβριο μέχρι την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου και ζητήσαμε να υπάρξουν και διαδικασίες επιπαραβάση αν χρειαστεί διότι όταν θα έχουμε κανόνες που δεν τηρούν κάποιοι ε, αν δεν ε, έχει αυτό κάποια συνέπεια θα δυσκολευτούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το Δουβλίνο έχει πεθάνει, μας το είπε και ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ δεν πιστεύω στην ιδέα ότι το πρόβλημα είναι ότι κάποιο άνοιξε τα σύνορά του. Όταν έχει σύνορα στη θάλασσα, δεν ανοίγει κάποια πόρτα. Είναι ανοιχτά από μόνο τους. Με τον κανονισμό του Δουβλίνου, Ιταλία και η Ελλάδα δεν είχαν κάποιο συμφέρον να φέρουν τους ανθρώπους αυτούς, δεν είχαν τρόπο να σταματήσουν αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους να έρθουν σε πιο ασφαλή εδάφη όπου ήταν οι οικογένειές τους, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους πολέμους, από την κλιματική αλλαγή ή από την απελπιστική κατάσταση στην οποία ζούσαν. Εκεί θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λοιπόν, να μεταρρυθμίσουμε το Δουβλίνο, να δούμε τι θα κάνουμε με τις νόμιμες και ασφαλείς οδούς πρόσβασης ε, για να τους βγάλουμε από τα χέρια αυτούς τους ανθρώπους των διακινητών αλλά για να βοηθήσουμε και αυτού του ανθρώπου που προσπαθούν να ξεφύγουν από του πολέμου και από την κλιματική αλλαγή. Και γι' αυτό απαιτούμε ευρωπαϊκέ πολιτικέ με μεγαλύτερη συνοχή, με καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και να σα δώσω, να σα πω και κάτι τελευταίο. Θα ξέρετε ότι οι αφρικανικέ χώρε τα τελευταία 50 χρόνια έχουν χάσει μέχρι λέγεται ένα τρισεκατομμύριο δολάρια έχουν χάσει λόγω της φοροδιαφυγής εταιριών και δικών μας Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο κόσμος για τον οποίο φεύγει ο κόσμος δεν είναι τόσο άσχετο με εμά από ό,τι νομίζουμε. Είναι πολιτικοί λόγοι, αποτελέσματα της δικής μας εξωτερικής εμπορικής πολιτικής που υποβαθμίζει τις χώρες αυτές, δημιουργώντας ανισότητες, αυξάνοντας ανισότητες στην κατανομή των πόρων, και των ε, δημοσιονομικών πολιτικών που έχουν ως αποτέλεσμα ότι εμείς με το ένα χέρι παίρνουμε αυτό που δίνουμε με την πολιτική ε, συνεργασία από την άλλη. Ευχαριστώ. Οπότε υπάρχει, μένα πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λάμπερτ. Ε, τα συμπεράσματα. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που ελέγχθησαν και είναι αλήθεια ότι ε, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, μας υπόθηκε προηγουμένως, δεν είναι μόνο, μόνο η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, είναι και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη στο παρελθόν, το 2015, είχε, είχαν φτάσει σε συμφωνία για το τι θα έκαναν σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση. Συμφώνησαν οι Υπουργοί Εσωτερικών. Και οι Πρωθυπουργοί τους τους είπαν ότι δεν μπορούν να το εφαρμόσουν σε κάποια κράτη-μέλη. Είχαμε δηλαδή έκτοτε αυτή την απόκληση. Το κρίσιμο εδώ, όταν μιλάμε για την αποτυχία του Δουβλίνου, είναι ότι η δομή του Δουβλίνου δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν έχουμε μια σημαντική ροή ανθρώπων. Μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό το πλαίσιο τη οδηγία προσωρινών ροών. Δεν συνέβη αυτό. Και τα κράτη-μέλη τελικά δημιούργησαν το ίδιο πρόβλημα το οποίο έχουν μπροστά του τώρα. Εάν δούμε ε, στη Μάλτα και στην Ιταλία ε, αυτά που ελέγχθησαν για την διάσωση στη θάλασσα, όπου είδαμε ανθρώπου να τους αφήνουν στη θάλασσα να πνιγούν επειδή οι ψαράδες φοβήθηκαν ότι εάν τους βοηθήσουν θα, διώ, θα υποστούν διώξεις. Ε, δεν υπήρχε συμφωνία για το τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια περίπτωση. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτική αποτυχία. Είναι και σε επίπεδο διαχείρισης αποτυχία. Και βεβαίως είναι κάτι σοκαριστικό. Οδήγησε σε τόσους θανάτους για ένα σύστημα ε, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κάλλιστα να οργανώσει και να λειτουργήσει. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ως μια από τις πιο πλούσιες περιοχές του κόσμου, ενώ είναι απίστευτο το τι κάνουν άλλοι, ε, ε τι να πω, να μην, ε, να μην κάνουμε καν προσπάθεια. Δεν λέω αυτό βέβαια στην πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα μοιράζει τις ευθύνε, το οποίο θα αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με ψυχραιμία, θα αναγνωρίζει ότι μας αφορά όλους, ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε, το οποίο δεν πρόκειται να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει απώλεια της ταυτότητας, της Ένωσης ε, για κανέναν, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τώρα για το πότε η θεωρία θα γίνει πραγματικότητα και το Δουβλίνο. Ακούστε, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και τώρα, χωρίς την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Και ένα από τα σημεία κλειδιά που πρέπει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά είναι η οικογενειακή επανένωση. Αυτό είναι κάτι επί του οποίου τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα. Αυτή τη στιγμή μαζί με μια οργάνωση που ονομάζεται Safe Passage, ασφαλής διέλευση, ε, κάνουμε μια δουλειά. Ε, είναι μια οργάνωση που αφορά κυρίως τις, την, τα περάσμα, το πέρασμα από Γαλλία στο Μένο Βασίλειο. Ε, η Βρετανική κυβέρνηση τώρα βέβαια ξέρετε ποια είναι, ας μην πω τίποτα. Αν δείτε όμως τη δουλειά που κάνει αυτή η οργάνωση Safe Passage στην Ελλάδα, θα σα πούν ότι εάν δεν παρέμουν σε μια υπόθεση οικογενειακή επανένωση μεταξύ ελληνικών αρχών και ενό άλλου κράτου μέλους, κατά 90% δεν συμβεί τίποτα. Όταν επεμβαίνουν, όταν κάνουν μέρο τη δουλειά, έρχονται σε επαφή με τα μέλη τη οικογένεια, τσεκάρουν κατά πόσο βρίσκονται όντω εκεί, κατά πόσο μπορούν όντω να δεχθούν έναν ασυνόδευτο ανήλικο, τότε σε 90% των περιπτώσεων αυτό λειτουργεί. Τι μου λέει αυτό, ότι όταν υπάρχει βούληση να κάνει κάποιο την προσπάθεια να διαθέσει του πόρου, τα χρήματα και να βοηθήσει του ανθρώπου αυτού, τα πράγματα πάνε πολύ πιο γρήγορα. Και αναθεώρηση της, αναμένως μάλλον στην αναθεώρηση του Δουβλίνου, ε, να κάνουμε τουλάχιστον ένα βήμα και να μην περιμένουν παιδιά για μήνε μέχρι να, βρουν μια οικογένεια και ενδεχομένω στο διάστημα, στο αυτό να χάσουν τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές. Ήταν μια εξαιρετικά ειλικρινή συζήτηση και γαλήνια ταυτόχρονα, ε, νυφάλια. Οι ευρωβουλευτές είναι στη διάθεσή σας βεβαίως για οποιαδήποτε ερώτηση. Μπορείτε να τους γράψετε μέσω mail. Σας ευχαριστώ όλους. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο, στο τελευταίο κομμάτι του προγράμματός μας και θα καλέσω την Σόφη Μαγκίνες σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας Η Σόφη είναι η επικεφαλής ε, της Μονάδας Πολιτικής και Νομικής Υποστήριξης της είπα αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών μπορείτε να κάτσετε εδώ Πριν ήταν μαζί μας και πριν σε ένα άλλο σεμινάριο πριν από κάποιο καιρό τα προηγούμενα ερωτήματά σας και αυτά που είπαν οι ευρωβουλευτές ε, στις απαντήσεις τους ε, δείχνει και πόσο το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια αυτό αποτυπώνει και το ότι ε, είναι ένα θέμα το οποίο ε, το βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς και έχει να κάνει με την ε, ανικανότητα τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάτι γι' αυτό είναι κάτι το οποίο διαφαίνεται στην σημερινή συζήτηση. Φαντάζομαι θα μιλήσετε για την προστασία των προσφύγων ε, υπό το πρίσμα της παραστατμοστίας. Γνωρίζετε βέβαια αυτή τη συζήτηση. Ε, έχετε μιλήσει με, την εισηγήτρια, μιλάτε συχνά με μέλη του Επικού Ίσως ε, μιας και βρίσκονται εδώ τόσοι δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη, ε, θα ήταν καλό να πούμε δύο λόγια για το τι κάνει η πατιαρμοστία και ποια είναι η άποψη της πατιαρμοστίας ό,τι αφορά την θεώρηση του κόσμου του Δουβλίνου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much and good afternoon. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα ήθελα στο όνομα της ΥΠΑ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μας δίνουν αυτήν την μοναδική ευκαιρία. Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία για μας να συνομιλήσουμε μαζί σας τους δημοσιογράφους από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να μοιραστούμε μαζί σας ε, κάποιες πληροφορίες ε, σχετικά με τις προοπτικές μας και κάποια βασικά μηνύματα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τα θέματα ασύλου και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ισχυρά και υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των ε, προσφύγων είναι πολύπλοκα και ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ποιοι είναι οι πρόσφυγες και πώς μπορούν να, να συνεισφέρουν θετικά στις ε, κοινωνίες που τους υποδέχονται. Επίσης, ε, συχνά στα ρεπορτάζ ε, υπάρχουν αναφορές που δυσκολεύουν την ζωή αυτών που προσπαθούν να προστατεύσουν τους πρόσφυγες, σπέροντας τον φόβο δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε στο προηγούμενο τμήμα της συζήτησης, ότι η κρίση το 2015 και 2016 ήταν σε μεγάλο βαθμό κρίση που δημιουργήθηκε από τα κράτη. Ήταν αποτυχία διαχείρισης και θέσπισης μηχανισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων προσφύγων και ασύλου. Θέλουμε λοιπόν ε, να σας βοηθήσουμε εσάς τους δημοσιογράφους να κάνετε τη δουλειά σας και να ε, σας μεταφέρουμε κάποια βασικά μηνύματα όσον αφορά την ε, δική μας προσέγγιση στην μεταρρύθμιση του ασύλου. Φυσικά έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ανεξάρτητες στατιστικές και αναφορές. Θα λάβετε ένα φυλάδιο με τους ε, συνδέσμους ε, προς ε, τις πηγές αυτές τις ανεξάρτητες. ελπίζω κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου να τα δείτε αυτά και στην οθόνη. Υπάρχουν λοιπόν διχτυακοί σπήλες, επιγραμμικές πηγές που μπορείτε να ελέγχετε σε καθημερινή βάση, στατιστικά σχετικά με τις αφήξεις από την Τουρκία προς την Ελλάδα που τώρα πια είναι πολύ περιορισμένες. Τα τελευταία ε, στοιχεία λοιπόν που έχει η πατιαρμοστία σας τα μοιράζουμε αυτή τη στιγμή ε, σε χαρτί. Επίσης ε, σας δίνουμε και τους συνδέσμους προς κάποιες από αυτές τις πηγές. Έτσι λοιπόν επιδεικνύουμε καλή βούληση και πειραζόμαστε μαζί σας σε τις πηγές που έχουμε. Όσον αφορά τα βασικά μηνύματά μας προς εσάς, θα ήθελα να πω ότι εμείς εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες εξετάζουμε την κατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κατά νου ότι 65 ε, ε, εκατομμύρια ανθρώπων αυτή τη στιγμή είναι εκτοπισμένοι ε, σε όλο τον κόσμο και πολύ μικρό ποσοστό αυτών βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τουρκία, το Λίβανο, τη Γιορδανία κλπ. Ενώ λοιπόν είδαμε το 2015 σημαντικές αφήξεις, οι αφήξεις αυτές έχουν πέσει πάρα πολύ το 2016 και φέτος και θα πρέπει να έχουμε κατά νου την κλίμακα του συνολικού προβλήματος. Όσον αφορά τους ετούντες άσυλο και τις ε, διαδικασίες ε, για την αίτηση διεθνούς προστασίας, πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες αυτές ε, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο καλύτερης διαχείρισης. Έχουμε υποβάλει μια σειρά προτάσεων για καλύτερη προστασία των προσφύγων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας δίνουμε τα στοιχεία ε, αλλά θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσο γίνεται καλύτερα τα στοιχεία. Αυτά που έχουν προταθεί για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρόταση στο μέλλον, και δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί ήδη τα ακούσατε, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Δουβλίνο 4, όταν θα καταφθάνουν ε, οι ε, πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ελέγχονται πρώτα για να διαπιστωθεί εάν μπορούν να εάν μπορούν να του υποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξεταστεί εάν υπάρχει άλλη χώρα με ασφαλείς διαδικασίες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες να μπορούν να μεταφερθούν. Στην πρόταση, λοιπόν, ε, έχουμε κάτι ανάλογο με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Ε, οι άνθρωποι καταφθάνουν από την Τουρκία, περνάνε από μια διαδικασία στην Ελλάδα και σε κάποιες περιπτώσεις μεταφέρονται πάλι πίσω στην Τουρκία. Από ό,τι γνωρίζουμε, κανένας σύρος δεν έχει επιστραφεί από την Ελλάδα στην Τουρκία, ε, σύμφωνα με τη συμφωνία αυτά, αυτή για κάποιους λόγους, για διάφορους λόγους. Η θέση μας εδώ είναι ότι πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα. Εξετάσαμε τις προτάσεις και εμείς προτείνουμε διαφορετική προσέγγιση. Προτείνουμε τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε οικογενειακή επανένωση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανθρώπου που καταφτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συγγενεί εδώ. Αυτοί που δικαιούνται η οικογενειακή επανένωση πάλι ε, θα μεταφέρονται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με τις προτάσεις που βλέπουμε εδώ πέρα και δεν ε, θα ε, έχουν δικαίωμα οικογενειακής επανένωση εντός Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμό αυτών που μεταφέρονται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, ε, θα μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ε, οι άνθρωποι όταν έχει, όταν ξεπερνάει ο αριθμός των αφιχθέντων το, κάποιον συγκεκριμένο αριθμό. Εμείς προτείνουμε σε κάθε κράτος μέλος όπου καταστάνουν ετούντες άσυλο να χρησιμοποιούνται, να εφαρμόζονται επιταχυμένες διαδικασίες ώστε γρήγορα να εντοπιστούν ε, αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία και να διαχωριστούν από αυτούς που δεν έχουν ανάγκη από προστασία. Για όσους ε, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ανάγκη προστασία ε, να προσφέρεται εθελοντική επιστροφή και αν δεν θέλουν να δεχτούν αυτήν την προσφορά και εφόσον δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος που να εμποδίζει την επιστροφή τους, να επιστρέφονται. Διότι με την παρούσα πρόταση θα γίνονται πολλές μετακινήσεις ανθρώπων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι πολύ δύσκολο να, το, να ελεγχθεί αυτό. Είμαι βέβαιη ότι ήδη σήμερα θα ακούσατε και θα γνωρίζετε τις πολιτικές συζητήσεις γύρω από την πρόταση για το Δουβλίνο. Δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχει συνένεση σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσετε. Και στην διάσκεψη της Νέας Υόρκης ε, του περσινού ε, Σεπτεμβρίου, οι ηγέτες του κόσμου ε, δεσμεύτηκαν με αλληλεγγύη και και μερισμό των ευθυνών να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Ε, με την νέα πρόταση του Δουβλίνου φαίνεται η ανάγκη αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να ε, αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να προσπαθήσουν να βρουν λύση μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου. Μία τελευταία παρατήρηση που ήθελα να κάνω έχει να κάνει με το φαινόμενο των δευτερογενών μετακινήσεων. Κάποιοι λοιπόν θα πούνε ότι άσχετα από το ποιες είναι οι διαδικασίες, ε, και πάλι θα μετακινείται κάποιος από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Καταλαβαίνουμε γιατί επιλέγουν κάποιοι να μετακινηθούν περαιτέρω. Συχνά αυτό έχει να κάνει με κακές ε, διαδικασίες ασύλου. Αυτή τη στιγμή τέσσερα κράτη-μέλη δεν πανούν καθόλου χρήματα στην ένταξη των ε, μεταναστών. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ε, ε, ένα πακέτο ε, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και μπορούν να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Τέσσερα κάτι μέλη δεν δαπανούν τίποτα στην ένταξη. Αν λοιπόν υπάρχει κράτος μέλος με πολύ χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων και δεν γίνονται επενδύσεις στην ένταξη, το σύστημα στη χώρα αυτή δεν διευκολύνει την οικογενειακή επανένωση ετούν τον άσυλο προς άλλες χώρες. Και αν παραμείνουν τα πράγματα έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα συνεχίσουν αυτές οι δευτερογενεί μετακινήσεις. Θέλουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα του Δουβλίνου και του επιμερισμού ε, των ευθυνών και τη αλληλεγγύης, εξετάζοντας τι λειτουργεί καλά και τι μπορεί να δώσει ε, πρόσβαση στην ε, προστασία για αυτού που την έχουν ανάγκη απομένει πάρα πολλή δουλειά να γίνει εξωτερικά, να δημιουργήσουμε συστήματα ασύλου και προστασίας σε άλλες χώρες. Ως οργανισμός δεν θεωρούμε ότι ο καθένας που έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας πρέπει να την βρει αυτή στην Ευρώπη. Θα πρέπει να οικοδομηθούν ανάλογα συστήματα στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες. Πρέπει να καλέσουμε τους εταίρους μας να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες και ε, όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση και την επανεκατάσταση. Στην διαφάνεια βλέπετε τους συνδέσμους προς κάποιες από τις πηγές πληροφόρησης που έχουμε. Ελπίζω όλοι σας ε, να έχετε λάβει ε, και σε χαρτί τις πληροφορίες αυτές και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες πηγές πληροφόρησης που έχουμε. Παρακαλώ δώστε μου ένα λεπτό ακόμα όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση ε, και την επανεκατάσταση με ιδιωτικές χορηγίες με υποτροφίες πανεπιστημίου για νέους, με ε, θεωρήσεις ε, δίνουμε πραγματικές εναλλακτικές λύσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Μέχρι τώρα όμως ε, οι δεσμεύσεις των κρατών μελών δεν έγιναν πίστευτες. Πέρσι είχαμε 8.000 ανθρώπους που ε, έλαβαν τέτοια μέτρα. Πρόπερσι ήταν 5.000. Κάποιος ε, λοιπόν ε, που προσπαθεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις νόμιμες οδούς για να αποφύγει τους επικίνδυνους τρόπους μετανάστευσης, εάν δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στα μέσα αυτά, ε, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Η διαχείριση τη μετανάστευση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή. Έχουμε υποβάλει προτάσει εφικτέ και σκόπιμε κατά τη γνώμη μα ε, και πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι για να, για διευκολυνθεί η νόμιμη μετανάστευση. Θα κλείσω εδώ για να σας δώσω χρόνο για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από αυτά που είπατε είναι ότι Ανεξάρτητα από τι θα συμβεί με αυτό το πακέτο μεταρρύθμισης ε, του συστήματος ασύλου, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή το να περάσει ο φάκελος τόσο στο κοινοβούλιο και να εγκριθεί δεν θα είναι πανάκια. Υπάρχουν άλλα ζητήματα, οι νόμιμες ε, οδοί εισόδου, η ε, ένταξη, υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία. Λοιπόν, ποιος θέλει ε, να θέσει ερωτήματα. Παρακαλώ. Σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομα μου είναι Άννα Καζαχαϊτον. είμαι freelance ε, δημοσιογράφος στη Φιλανδία. Το ερώτημά μου έχει να κάνει τις, ε, με τις σχέσεις μεταξύ της υπασταρμοστίας των ε, ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών κυβερνήσεων. Η εσεί σα πρόκειται κυρίω στι εθνικέ κυβερνήσει. Πόσο μπορείτε να του πιέσετε όμω και πόσο σα ακούν. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο ερώτημα. Γεια σα. Από την Πολωνία. Είπατε ότι υπάρχουν τέσσερι χώρε που δεν χρησιμοποιούν τον προπολογισμό για την ένταξη. Δεν διαθέτουν χρήματα για την ένταξη των μεταναστών και των ασύλου. Ποιε είναι αυτέ οι χώρε και γιατί είδου προπολογισμό μιλάμε, γιατί είδου κονδύλια μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Να ξεκινήσω με το ερώτημα από την Πολωνή δημοσιογράφο σε ό,τι αφορά τις χώρες που δεν διαθέτουν χρήματα στο ΆΜΙΦ. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες αυτές ε, και βεβαίως υπάρχει ειδικό διακανονισμός για την Ελλάδα διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα η Ελλάδα. Ζητούμε λοιπόν και από την Ελλάδα να διαθέσει χρήματα για την ένταξη, η Βουλγαρία επίσης. Ε, για την Πολωνία, από όσο ξέρω, έχουν δοθεί κάποια επιπλέον χρήματα για περαιτέρω χρηματοδότηση από το ΆΜΙΦ. Ε, αν έρθει σε επαφή μαζί μας μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία για, το, για τι είδους κονδύλια μιλάμε. Ε, τα χρήματα αυτά από το ΆΜΙΦ είναι κρίσιμα έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να τα χρησιμοποιήσουν ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, κανονικά είτε από το κράτος είτε από ΜΚΟ οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται σε, αυτά τα, σε αυτές τις χώρες ε, υποστήριξη γλωσσικής εκμάθησης, υποστήριξη σε ό,τι αφορά τι τις συνθήκες υποδοχής, διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης για να βοηθηθούν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες ε, διασπορές προσφύγων από κάποιες χώρες σε κάποια κράτη-μέλη. Βεβαίως, στο παρελθόν δεν υπήρχε καμία κοινότητα προσφύγων τον ασύλο εκτός Ευρώπης. Όλοι λοιπόν κάπου κάπου ξεκινάνε. Ε, και εδώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ε, και πολλές πληροφορίες για τις πρακτικές ένταξης που μπορούν να λειτουργήσουν και υπάρχει και χρηματοδότηση. Τώρα, αν ενδιαφέρεστε, μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία ε, για την κατάσταση αναχώρα. Σας ενθαρρύνω να ε, το αναζητήσετε αυτό για να δείτε αν δαπανώνται τα χρήματα, γιατί δεν δαπανώνται όταν δεν δαπανώνται, έτσι ώστε να υπάρξει μια ε, ενθάρρυνση προς τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά, να τα διαθέσουν. Υπάρχουν πολλές κοινότητες ε, στα κράτη-μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν σε διάφορα project ε, επιγραμμικά υπάρχουν κοινότητες που θέλουν να βοηθήσουν πρόσφυγες ε, μέσω δραστηριότητα στα σχολεία ή αλλού. Η χρηματοδότηση λοιπόν προς ΜΚΑ όμικρον ε, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Με αυτές τις τρεις γνωρίζω, δεν ξέρω ποια είναι η τέταρτη. Υπάρχει μια τέταρτη, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα και δεν θέλω βεβαίω να πω κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές σε ό,τι αφορά το ερώτημα από τη Φιλανδία, από τη Φιλανδία δημοσιογράφο, για τις σχέσεις με τα Εθνικά όργανα της Ένωσης, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ καλή ε, σταθερή σχέση σε επίπεδο είπα που ε, ο είπα συχνά είναι εδώ στην Ευρώπη ε, και μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Κομισιόν ε, καθημερινά ουσιαστικά είμαστε σε επαφή. Ε, συχνά μας, ζητά, ζητούν τα κράτη-μέλη της Ένωσης και τα θεσμικά όργανα να παράσχουμε ε, συμβουλές. Δεν είδα να υπάρχουν πάντως εμπόδια. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο έργο μας, είμαστε διαφανείς στις προτάσεις που υποβάλλουμε και πολλά κράτη-μέλη στην πραγματικότητα όλο και πιο συχνά απευθύνονται σε εμά για τέτοιου είδου συμβουλέ για το πώ να προχωρήσουν. Η Πατιαρμοστία έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτών, στο θέμα δηλαδή της ε, μαζικής μετακίνησης ατόμων ε, και είδαμε ότι υπάρχουν ε, έτσι ε, ότα από τα κράτη-μέλη και έχουμε βεβαίως εκφράσει και τις ανησυχίες μας και τις κριτικές μας όποτε αυτό ε, χρειάστηκε ε, και για τις εξελίξεις ε, που δεν μας αρέσουν βγάζουμε αναγνωθέντα τύπου ε, παίρνουν πρωτοβουλίες δηλαδή δεν μας περιορίζει κάποιος είμαστε μια διακυβερνητική οργάνωση και αυτή τη δουλειά θα τη συνεχίσουμε με σταθερότητα και διαφάνεια Ευχαριστούμε λοιπόν. Έχουμε χρόνο για άλλες δύο Δεν νομίζετε ότι με τις νέες ε, προτάσεις ε, και εφόσον υπάρξει κάποιο είδου δέσμευση για πιο εθελοντική κατανομή ε, με τα, βάσει των κειμένων του Δουβλίνου θεωρείτε ότι η επαναγκατάσταση ε, θα πάψει να λαμβάνει χώρα ε, στα κράτη-μέλη. Κάτι που αφορά εσάς ω είπατε των Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτό που έχει συμβεί με το μηχανισμό μετεγκατάσταση είναι δυστυχές. Διαρκώς κάνουμε εκκλήσει προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσει τους. Ορισμένα κράτη-μέλη το έχουν πράξει. Ένα έχει ε, τηρήσει πλήρω τι δεσμεύσει του, αλλά έχουν μείνει πίσω σαφώ. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί μεγάλε πιέσει. Θα ακούσετε και τον κύριο Αβραμόπουλο στη συνέχεια. Έχει πέσει πολύ η Κομισιόν. Θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε μετεγκαταστάσεις εθελοντικές ε, να παρέχουν εθελοντικά αλληλεγγύη. Αλλά έχουμε κάνει και έκκληση προς τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ τους ε, για επιμερισμό της ευθύνης και της αλληλεγγύης. Ο λόγος είναι ότι αναγνωρισμένα αυτή τη στιγμή υπάρχει δυσπιστία. Κάποια κράτη-μέλη δεν βασίζονται στις υποσχέσεις άλλων θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν δεσμευτικέ συμφωνίε που θα παρέχουν την απαραίτητη σαφήνεια. Όταν η κατάσταση αφορά 160.000 ανθρώπου, αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολο αν κάποιο έχει συνυπογράψει σε κάτι το οποίο έχει συγκεκριμένου χρόνου, αριθμού, δεσμεύσει, αντί να αφήνουμε τα πράγματα εθελοντικά. Αυτό που θέλουμε να πούμε στα κράτη-μέλη που εμφανίζουν δισταγμούς. Ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα αλλάξουν οι τάσεις. Ε, κάποια στιγμή μπορεί αυτά τα κράτη-μέλη να, χρησιμοποιη... να χρειάζονται άλλα κράτη-μέλη ε, για λόγους μετεγκατάστασης. Δεν είναι λοιπόν μόνο υποχρέωσή τους να βοηθήσουν τους ετούντες άσυλο και τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ε, συμφέρει και τα ίδια να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα αλληλεγγύης. Ναι, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον επιχείρημα και είναι η πρώτη φορά που το ακούμε σήμερα το μεσημέρι. Άλλες ερωτήσεις, τελευταίες ερωτήσεις. Yeah. No. Όχι. Παρακαλώ. Για να επανέλθω, μιλάω για την επανεγκατάσταση. Αυτή με ενδιαφέρει. Δεν, βρίσκει, δεν απειλείται σε περίπτωση που ε, δώσουμε περισσότερη προσοχή στην αντικατάσταση. Εννοείται όσον αφορά την επανένταξή τους. Ενώ ότι την επανεγκατάσταση. Α, το resettlement. Ναι, συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει. Λοιπόν, όσον αφορά την επανεγκατάσταση, ε, είναι στο ίδιο επίπεδο με την μετεγκατάσταση κατά την άποψή μας με την επανεγκατάσταση κάνουμε διαρκώς έκκληση στα κράτη-μέλη να μην παρουσιάζουν τα νούμερα της μετεγκατάστασης ως νούμερα επανεγκατάστασης κάναμε έκκληση προς τα κράτη-μέλη να μας δίνουν νούμερα εξαψήφια όσον αφορά την ε, επανεγκατάσταση. Η επανεγκατάσταση σημαίνει φυσικά ανθρώπων εκτός, από, ε, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πρόγραμμα μετεγκατάσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δημιουργήθηκε πριν λίγα χρόνια, αλλά οι αριθμοί δεν είναι μεγάλοι. Κάνουμε έκκληση λοιπόν προς τα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το πρόγραμμα των επανεγκαταστάσεων και να συνεχίσουμε με την κατάσταση. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ορισμένες ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο παρουσιάζουν το εξής επιχείρημα και το έχουν παρουσιάσει και ορισμένα μέσα μαζική ενημέρωση ότι η οικογενειακή μεταγκατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει ε, παράγοντα έλξης προς την Ευρώπη. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Η οικογενειακή επανένωση δηλαδή συγγενείς που έρχονται ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζεται από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και μέσω διαφόρων ε, εθνικο, διεθνών μέσων και μέσω της οδηγίας, της οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα. Για το επιχείρημα αυτό και για το παράγοντα έλξης που ακούμε συχνά ε, όταν προσπαθούμε να προωθήσουμε την νόμιμη κίνηση ανθρώπων, πρέπει να πω το εξή. Εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμοι τρόποι οικογενειακής επανένωσης, ε, οι άνθρωποι θα προτιμούν επικίνδυνες οδούς ε, για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε τέτοιο κίνδυνο χωρίς να έχουμε ε, αποδεικτικά στοιχεία, αλλά πιστεύουμε ότι πολλοί κόσμος ε, κινείται για αυτό το λόγο παράνομα. Οπότε συμφέρει τα κράτη-μέλη να διοργανώσουν πιο καλύτερα τις νόμιμες μετακινήσεις. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την οικογενειακή επανένωση είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, όταν έχουμε οικογένειες ε, διασπασμένες, έναν γονέα χωρίς παιδί, παιδί χωρίς γονείς ή αδέρφια, ε, είναι πολύ δύσκολη η ένταξή τους ε, στο κράτος μέλος όπου βρίσκονται. Πολλά κράτη-μέλη ανησυχούν για την ένταξη, για τον κοινωνικό ιστό των δικών τους κοινωνιών, ε, σε περίπτωση μη ένταξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Οπότε, κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να ενταθεί η έλξη, ουσιαστικά όταν δεν επιτρέπουμε την οικογενειακή επανένωση, υποσκάπτουμε την ικανότητα ένταξη των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποτελεί βασικό κίνδυνο, πιστεύω, που ανισχύει τα κράτη-μέλη. Επίση, να υπογραμμίσω το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή η οικογενειακή επανένωση για ανθρώπου που έρχονται έξω, εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σχεδόν αδύνατη. σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος ε, πολίτη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε μια πρεσβεία, συμπληρώνει ένα σωρό χαρτιά, κάνει αίτηση για θεώρηση, πρέπει να εγκριθεί η θεώρηση, πρέπει να πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα, να αποδείξει του οικογενειακού δεσμού, τα εμπόδια. Είναι τεράστια. Και προσπαθούμε να συνεργαστούμε με ΜΚΟ και άλλου ε, για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν λειτουργεί καθόλου και με την οικογενειακή επανένωση πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα. Το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών ε, να επανενωθούν με τις οικογένειέ τους χωρίς να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια και επίση να δώσουμε τη δυνατότητα σε οικογένειε και σε ενήλικε να ενταχθούν καλύτερα στα κράτη-μέλη που βρίσκονται. Μια τελευταία ερώτηση από πλευρά μου. Προφανώς ε, ε, γίνεται μια πολιτική μάχη εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών όπως ακούσαμε προηγουμένως. Από τη δική σας επαφή με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τα δύο θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείτε ότι είναι πιθανό να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία επένως Είστε επιφυλακτικοί, είστε αισιόδοξοι. Είναι δύσκολο να πει κανείς πότε θα επιτευχθεί η συνένεση αλλά δεν βλέπουμε για ποιο λόγο να μην επιτευχθεί. Τα προβλήματα δεν είναι τόσο περίπλοκα που να μην είναι δυνατή η επιτεύξη μια συμφωνία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα καταλήξουν σε μια λύση. Πολλά από τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν νόημα φυσικά απολύτως πολλές παρατηρήσεις ε, για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το Δουβλίνο είναι ρεαλιστικά. Οι πολιτικοί τώρα θα πρέπει να δουν κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθούν συμφωνίες. Αλλά εμείς ελπίζουμε ότι αν αποδειχθεί ότι λειτουργεί κάπως καλύτερα με την κατάσταση και αυξάνονται οι αριθμοί και αν ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι του συμφέρει η σωστή διαχείριση τη μετακατάσταση, τότε πιστεύουμε ότι θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων αυτών. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε ότι είναι δυνατή η διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Έχουμε στείλει συγκεκριμένε προτάσει για το πώ μπορεί να γίνει αυτό και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεωρούν τον εαυτό του ω χώρε που έχουν να παίξουν κάποιο ρόλο. Να αποφύγουμε αυτή την ορολογία του που εξακολουθούμε να ακούμε για ετούντες ασύλους που, ασύλου που έχουν μείνει κολλημένοι σε κάποιες χώρες ε, ή σε κάποιες χώρες διέλευσης. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να έχουν ε, συστήματα ασύλου και ένταξης που να λειτουργούν. Αν έκανε μια μικρή προσπάθεια κάθε κρατός μέλος, θα μπορούσε, πιστεύουμε, να επιτευχθεί κάποια πολιτική συνένεση. Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ διαφωτιστικές σας ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας όλα τα στοιχεία, τις πηγές, τα στατιστικά στοιχεία που μας βοηθούν, βοηθούν τους δημοσιογράφους ε, στη δουλειά τους. Ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη σήμερα είναι ο Επίτροπος κύριος Αβραμόπουλος. Μου είπαν ότι έφυγε από το κτίριο Μπερλεμό πριν από λίγα λεπτά οπότε θα πρέπει να είναι σύντομα κοντά μας. Εγώ θα φύγω για μια μικρή ανάγκη από την αίθουσα. Μην φύγετε, ώστε να είμαστε όλοι εδώ όταν έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής συνεδρίασης. Και μετά θα ακολουθήσει μία ώρα και 15 λεπτά για οτιδήποτε επιθυμείτε να κάνουμε και μετά αν θέλετε μπορείτε να έρθετε στο κοκτέιλ δικτύωση, που ξεκινά στις 6. So just uh, to announce that... Uh, Να σας ενημερώσω. Υπάρχει μια καθυστέρηση από την Επίτροπο, αλλά δεν θα αργήσει. Μην αποθαρρύνεστε. Uh, Παρακαλώ πάτε θέσεις κυρίες και κύριοι. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, τον κύριο Βραμόπουλο την κυρία Βίξτρομ βεβαίως, την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας. Ε, να σας πω ότι σήμερα το πρωί διάβασα πριν τα γενέθλιά σας, οπότε χρόνια πολλά. Θα ήθελα να μιλήσω για την πρόταση ενό κοινού συστήματο ασύλου στην Ευρώπη. Είναι μια πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν πριν από μερικού μήνε. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, το παρακολουθείτε βεβαίω το ζήτημα, παρακολουθείτε τι γίνεται εδώ και το τι γίνεται σε επίπεδο Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εγώ δεν θα σχολιάσω τι γίνεται εκεί. Ε, Πάντως χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άργησα λίγο διότι είχα μια συνάντηση με τον ε, αντιπρόεδρο της Ακτής Λεφαντοστού που κράτησε λίγο περισσότερο για προφανείς λόγους. Ε, είμαι πάντως εδώ μαζί σας ε, για να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις σήμερα το απόγευμα, να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε. Γι' αυτό το εξαιρετικά, εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Χαίρομαι επίση ιδιαίτερα που είναι εδώ η Σεσέλια Βίξτρομ, ε, η οποία μου ζητάει να μιλήσω ελληνικά. Είναι από τους ευρωβουλευτές η κυρία Βίξτρομ που γνωρίζει η μητρική μου γλώσσα τα ελληνικά, η Σουηδή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σεμινάριο, όπως αντιληφθήκατε. Πολλές πληροφορίες ε, θα λάβετε και βεβαίως θα φωτίσει τις πληροφορίες αυτές κάποια από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με το Λονδίνο και τον Ηνωμένο Βασίλειο ε, για την ε, φρικτή επίθεση που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ ε, την αστυνομία του Λονδίνου και τις αρχές αποβολής του νόμου για την εξαιρετικά γρήγορη και αποτελεσματική αντίδρασή τους. Ξέρουμε όλοι ότι η τρομοκρατία μας επηρεάζει όλους το ίδιο. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και δυνατή στην κοινή μας απάντηση. Είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Καθώς συζητούμε τα ζητήματα ασύλου σήμερα, θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ τρομοκρατίας και μετανάστευσης ή μεταξύ τρομοκρατών και τούντων άσυλο. Ακούμε φωνές που δεν θέλουν να δεχτούν ετούντες άσυλο για λόγους ασφαλείας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς την, από την τρομοκρατία φεύγουν. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ετούντες άσυλο εμπλέκονται σε ζητήματα ασφάλειας. Η επίθεση στο Βερολίνο είναι ακόμα φρέσκια στη μνήμη μας. Πρέπει να επαγρυπνούμε και είμαστε και επαγρυπνούμε. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε αυτήν την ψευδή ρητορική που ε, τσουβαλιάζει τους μετανάστες, τους πρόσφυγες ε, και τους τρομοκράτες. Έτσι είναι να δεχόμαστε αυτή την αφήγηση της ε, διέρεσης και τη αντιπαράθεσης που προωθούν τρομοκράτες. Όπως ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κοινό σύστημα ασύλου το οποίο να μπορεί να αντέχει στο μέλλον, να βασίζεται σε κοινού κανόνες και μία ίση κατανομή ευθυνών. ισομερή καταμερισμό ευθυνών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ανοιχτή και επικοδομητική συζήτηση όχι μόνο με τους νομοθέτες αλλά και με το κοινό. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες ε, των συμπολιτών μας και των κοινοτήτων μας θα αντιμετωπιστούν μέσω της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έχουμε μπει σε μια εποχή κινητικότητας των ανθρώπων. Το θέμα δεν είναι λοιπόν πώς θα σταματήσουμε τη μετανάστευση. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε. Η κρίση των προσφύγων μας έμαθε ότι τα αμυγός εθνικά μέτρα δεν δίνουν ικανοποιητικές λύσεις για κανένα κράτος μέλος ξεχωριστά και βεβαίω ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Μια προσέγγιση κατακρεματισμένη, εσωστρεφής, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της, με, της, της μετανάστευσης ε, σφαιρικά, αλλά ε, υπονομεύει το ίδιο το ευρωπαϊκό σχέδιο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση σε ένα πνεύμα πραγματικής αλληλεγγύης και ευθύνης. Είτε για να βελτιώσουμε την επιστροφ, τις επιστροφές, την αντιμετώπιση ε, των ε, διακινητών και τη θωράκη των συνόρων. Κανεί δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνο του. Καμία χώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να προστατέψουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να επιτρέψουμε στο σύστημα ασύλου να προσφέρει προστασία για αυτούς που τη χρειάζονται, για να μπορέσουμε ε, να ε, εξαρθρώσουμε τα δίκτυα των διακινητών και να τους διώξουμε και βεβαίως ε, αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σφαιρική προσέγγιση στην διαχείριση της μετανάστευσης. Περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει να αφαιρέσουμε ευθύνε ή αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη όπως κάποιοι φοβούνται. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει μια καλύτερη κοινή διαχείριση απέναντι στην κοινή πρόκληση πολλές κοινέ δράσεις έχουν συμφωνηθεί, σημαντικές κοινέ δράσεις, δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται. Η προσέγγιση των hot spot, τα, συστήματα, τα, τα προγράμματα μεταγκατάστασης και επαναγκατάστασης, η προσπάθεια επιστροφής των παράτυπων μεταναστών και η αυξημένη συνεργασία με τρίτες χώρες για τα ζητήματα επανεισδοχής. Δεν αρκούν όμως αυτές οι δράσεις. Για να ολοκληρώσουμε τη συνολική μας προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, η μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου είναι ένα, μια απαραίτητη προϋπόθεση. Εάν η κρίση των προσφύγων των περασμένων τριών ετών μας έδειξε ένα πράγμα, αυτό είναι ότι το status quo του κοινού συστήματος ασύλου δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Οι δομικές αδυναμίες στο παρόν σύστημα κατέστησαν προφανείς με την κρίση αυτή. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ασύλου. Οι συνθήκες υποδοχής των ετούντων, τα ποσοστά αναγνώρισης, και ο τύπος προστασίας που χορηγείται ε, για τους δικαιούχους πλήθους προστασίας ποικίλουν. Αυτές οι διαφορές είναι που οδηγούν στις δευτερογενείς μετακινήσεις και στο asylum shopping. Και αυτό οδηγεί σε μια ανισομερή κατανομή των ευθυνών μεταξύ κρατών μελών για να μπορέσει να δοθεί προστασία σε αυτούς που τη χρειάζονται. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα ισχυρό σύστημα ασύλου, ένα σύστημα που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην ίση κατανομή ε, ευθυνών. Ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να αντέχει στις κρίσεις αλλά ταυτόχρονα να είναι δίκαιο. Χρειαζόμαστε δομές και εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα σύστημα το οποίο να αντέχει στο μέλλον όπου κανένα κράτος μέλος να μην μένει μόνο για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα μόνο του. Για το σκοπό αυτό, τα εθνικά συστήματα ασύλου πρέπει να έρθουν πιο κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά επίσης ε, θα μειώσει τα κίνητρα για την αναζήτηση ευνοϊκότερου καθεστώτος ασύλου ή της κατάχρησης ε, από τους ετούντες. Η αμοιβή εμπιστοσύνη είναι κάτι απαραίτητο όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, διασφαλίζει επίσης η ίση αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ετούντων άσυλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προτείνουμε να ενσωματώσουμε στο σύστημα διάφορα στοιχεία τα οποία θα βελτιώσουν την ευρωπαϊκή ένταξη. Αυτό θα γίνει μέσω μεγάλης αναρμόνισης, ευρύτερης σύγκλησης ε, της αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σύστημα ίσης ε, κατανομής των ε, αιτούντων άσυλων μεταξύ των κρατών μελών. Το πακέτο μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής προτείνει ένα σύστημα όπου οι διαδικασίες και τα χρονοδιάγραμματα θα έχουν βελτιωθεί, όπου τα δικαιώματα των ετούντων ε, θα διασφαλίζονται σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών και όπου τα κριτήρια ε, λήψης διεθνούς προστασίας θα έχουν αναρμονιστεί ακόμη περισσότερο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ετούντες θα την χάνουν ίσης ε, μεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση βάσει συγκεκριμένων προτύπων. Επίση, αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα των δευτερογενών μετακινήσεων. Προτείνουμε λοιπόν την εφαρμογή των ε, αναλογικών κυρώσεων όσον αφορά τις ε, συνθήκες ε, διαδικασιών και υποδοχής όταν οι ετούντες δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η επιτυχία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεγγύη. Η γεωγραφική θέση δεν μπορεί να ορίζει το βαθμό υπευθυνότητα, το βαθμό ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δυσανάλογο φόρτο σε κάποια κράτη-μέλη που τυχαίνει να βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή μα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ουσιώδου σημασία. Γι' αυτό το σκοπό προτείνουμε να έχουμε έναν διορθωτικό μηχανισμό ε, κατανομής ε, ενσωματωμένο στο νέο σύστημα του Δουβλίνου. Το να προστατεύουμε την, ε, μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα χρειαζόμαστε ένα σύστημα Δουβλίνου σαφές, προβλέψιμο, αποτελεσματικό και δίκαιο. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε δέσμευση από τα κράτη-μέλη. Κάτι που μεταφράζεται σε σαφείς και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ε, σε μελλοντικές κρίσεις να υπάρχει καταμερισμός της ευθύνη και αναδιανομή της. Όταν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη ε, υφίστανται υπερβολικό φόρτο. Σκοπός μας ε, είναι επίσης να αποθαρρύνουμε τις ανεξέλεγκτες ε, παράτυπες μετακινήσεις, να παρέχουμε οργανωμένους και ασφαλείς ε, οδούς προς την Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε και ένα ενωσιακό πλαίσιο επανεγκατάστασης που θα ε, δημιουργεί μια κοινή προσέγγιση ασφαλείς νόμιμες οδούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ένα ενωσιακό πλαίσιο η επανεγκατάσταση θα μειώσει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών πρακτικών. Επίσης θα θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ισχυρότερη θέση διεθνώς θα της δώσει τη δυνατότητα να μιλάει με μία φωνή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πείσουμε καλύτερα τους διεθνείς μας εταίρους να αναλάβουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο ευθύνης. διότι η εξωτερική και εσωτερική διάσταση της διαχείρισης ε, της μετανάστευσης ε, είναι αλληλένδετες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εντείνει τη δεσμευσή μας με κάποιες τρίτες χώρες κλειδιά για να αντιμετωπίσουμε τις ε, βασικές αιτίες της μετανάστευσης, για να βελτιώσουμε τις καταστάσεις της χώρας καταγωγής και διέλευσης, για να καταπολεμήσουμε τους διακινητές, να βελτιώσουμε τους επαναπατρισμούς και να ενισχύσουμε τις νόμιμες οδούς. Σε αυτό ακριβώς επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις μου πριν από 25 λεπτά με τον ε, Αντιπρόεδρο της Ακτής Ελεφαντοστού και με πολλούς άλλους αρχηγούς που μας επισκέπτονται σήμερα. Αυτό πηγαίνει παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, για να φέρουν αποτελέσματα οι δρέσεις μας, ε, έχει έρθει η ώρα τα κράτη-μέλη να δείξουν την πολιτική τους ε, δέσμευση και βούληση ώστε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ειδικότερα του συστήματος του Δουβλίνου. Τα κράτη-μέλη καθώς και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ε, η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου να είναι φιλόδοξη. Θα πρέπει να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα μπροστά ε, από άποψη αποτελεσματικότητα, σύγκλησης, καταπολέμησης των δευτερογενών μετακινήσεων και αλληλεγγύης. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, Εστονική Προεδρία που αναλαμβάνει αρχές Ιουλίου να συνεχίσουν τις ακούραστες προσπάθειες της Μαλτέζικης Προεδρίας ώστε να επιτευχθεί συμβιβασμός με όλα τα κράτη-μέλη επί ενός μηχανισμού αλληλεγγύης που θα είναι προβλέψιμος και που θα ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αφήνεται μόνο του. Επίσης υπολογίζουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στα διάφορα ε, θέματα που εξετάζει και δράτω με τις ευκαιρίες ε, που βρίσκεται εδώ η Σεσίλια για να σας πω ότι από την αρχή πριν από αρκετά χρόνια ο κύριος υποστηρικτής των προσπαθειών μας όλων των πρωτοβουλίων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή υπήρξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί φίλοι, το φαινόμενο της μετανάστευσης πρέπει να το δούμε με ένα στρατηγικό, ολοκληρωμένο και θετικό τρόπο. Όπως είπα νωρίτερα, η κινητικότητα και η μετανάστευση είναι χαρακτηριστικά του σημερινού κόσμου. τις προκλήσεις θα πρέπει να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης εξαρτάται από όλους εμάς να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αβραμόπουλε. Θα ακούσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις. Παρακαλώ, υπάρχει κάποιος που δεν έχει θέσει ερώτηση μέχρι τώρα. Ο κύριος εδώ, η κυρία και εσείς εκεί πίσω. Παρακαλώ. Λέγομαι τη Σίλερ 4 από την Ουγγαρία. Η κυρία Βίκστρομ ανέφερε νωρίτερα ότι κατά τη γνώμη της πάγωμα των διαφορετικών ταμείων θα μπορούσε να επιβληθεί ως κύρωση στις χώρες που δεν δέχονται ετούντες άσυλο. Αντίθετα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιείχε πρόστιμο ανά ετούντα άσυλο. Ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό. Πιστεύετε ότι από νομικής πλευράς είναι εφικτό κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του ισχύοντος πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, νομίζω καλύτερα είναι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις μία προς μία. Ε, προέρχεστε από μία κεντρική και μία από τις πιο ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Οι πρόγονοί σας γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να είναι κανείς πρόσφυγας. Το 1958 πάνω από μισό εκατομμύριο ε, Ούγγροι ε, έφυγαν από την Ουγγαρία. Ναι, αλήθεια, θα περιμέναμε περισσότερα από την Ουγγαρία. Και θα περιμέναμε, ακόμα περιμένουμε, η Ουγγρική κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτά που συμφωνήσαμε όλοι πριν δύο χρόνια στο Λουξεμβούργο. Όπως είπε στην αρχή, είναι η ώρα να επιδείξουν όλα τα κράτη-μέλη ευθύνη και αλληλεγγύη. Αυτά δεν είναι απλά λόγια. Η ευθύνη και η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο όροι ηθικής. Είναι και νομικοί όροι. Ε, συμπεριλαμβάνονται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από την αρχή. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν για όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν την πολιτική που έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Το μήνυμα λοιπόν είναι πολύ σαφές. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που έχω πει στο παρελθόν και που είπα ήδη σήμερα το πρωί. Ναι. Θα ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση. Πιστέψτε με, αυτό δεν με κάνει ευτυχή. Αλλά πρέπει να το κάνω. Διότι αυτός είναι ο ρόλος ενός επιτρόπου, να υπερασπίζεται τις συνθήκες. Από την άλλη, πιστεύω ότι είναι πολιτική, ηθική και νομική υποχρέωση στο όνομα... Ε, ε, ε, όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν όλα όσα έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Διότι η μεταναστευτική κρίση και το υπονόησα αυτό στην αρχή της ομιλίας μου, ε, θέτει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και ίσως αυτό να ακούγεται ε, υπερβολή. Αλλά πιο πολύ από την οικονομική κρίση, η μεταναστευτική κρίση θέτει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό όραμα, το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και έχουμε πολιτικό, ιστορικό, ηθικό χρέος να προστατεύσουμε αυτά που κληρονομήσαμε και να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την ενότητα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, yes, hello. My name is Γεια σας, Σοφιτρίνεν από την Φινλανδία. Εκπροσωπώ ημερήσια εφημερίδα. Είπατε ότι ο στόχος ε, είναι να ε, υπάρξουν νόμοι οδοί προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη έχουν καταστήσει πιο δύσκολο να εισέλθει κανεί στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επανένωση έχει γίνει πιο δύσκολη στη Φιλανδία, για παράδειγμα, διότι έχει θεωρηθεί παράγοντας προσέλκυσης. Με τι συγκεκριμένου τρόπους θα ενθαρρύνεται τα κράτη-μέλη να ανοίξουν περισσότερες νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη. Ο κύριος αυτή είναι η στρατηγική μας, να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς για αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε κάποια χρόνια από τώρα η Ευρώπη θα έχει ανάγκη από εργατικό δυναμικό. Θα έχει ανάγκη τους μετανάστες. Όπως πολύ σωστά είπατε όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νόμιμες διόδους. Όταν αυτή η κρίση χτύπησε την πόρτα της Ευρώπης, ε, η Ευρώπη ε, βρέθηκε προ μεγάλης έκπληξης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τα κράτη-μέλη είχαν εμπειρία διαχείρισης ενός τέτοιου φαινομένου. Δεν βρισκόμαστε όμως πια εκεί που βρισκόμασταν πριν δύο χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Έχουμε λάβει πολύ σημαντικές ε, αποφάσεις, έχουμε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι άλλο απρόβλεπτο σε αυτήν ε, την αποσταθεροποιημένη περιοχή από την οποία προέρχονται όλοι αυτοί οι μετανάστες. Όπως είπα και πριν όμως, δημιουργήσαμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, υιοθετήσαμε νέα νομοθεσία, ώστε όσοι θέλουν να εισέλθουν στην Ευρώπη ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες, να ε, τους υποδεχόμαστε και να τους καλωσορίζουμε εδώ. Πρέπει όμως να είμαστε απόλυτα σαφείς όσον αφορά κάτι άλλο. Όσοι έχουν ήδη καταφτάσει στην Ευρώπη, παράνομα, κάποιους τους εκμεταλλεύτηκαν ε, διακινητές. Αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Γι' αυτό ανέφερα κατά την εισαγωγή μου ότι ασχολούμαστε με την ε, επανεισδοχή και τις επιστροφές. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερη. Να σας θυμίσω, όπως είπα ήδη στην αρχή, ότι έχουμε προτείνει ευρωπαϊκό ε, σύστημα επανεγκατάστασης. Γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν πάνω στο θέμα αυτό. Τελευταία ερώτηση, κατόπιν θα πρέπει να κλείσουμε, διότι ο Επίτροπος... Όχι, όχι, μην κατηγορείτε τον Επίτροπο, διακόπτει ο Επίτροπος, εγώ μπορώ να κάτσω εδώ μέχρι αύριο. Όχι, όχι, καθυστέρησα, οπότε μπορώ να κάτσω λίγο παραπάνω. Από τη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς βλέπει την ε, αντιμετώπιση της Βουλγαρίας. Τι, λέτε, τον αγώνα της Βουλγαρίας κατά των ε, προσφύγων, ε, λέει ο, ο Επίτροπος η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς αξιολογεί τις πολιτικές της Βουλγαρίας. Και ο Βούλγαρος Πρόεδρος, ο κ. Ράτεφ, ζήτησε μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να δώσει χρηματοδότηση τέτοιου ύψους. Αγαπητέ φίλε, ήδη το κάναμε. Την Βουλγαρία τη στηρίζουμε πρακτικά, πολιτικά και οικονομικά. Στηρίζουμε τη Βουλγαρία ήδη από την αρχή. Είχα συζήτηση πριν 6 μήνες με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Μπόρισεφ, που επανεξελέγει πάνω στο θέμα αυτό. Πρόσφατα, η Βουλγαρία βρέθηκε υποπίεση, διότι δεδομένου του ότι η δήλωση Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί και επειδή έχει κλείσει ο διάδρομος Μπουρκάς, οι μετανάστες έχουν επιλέξει άλλες οδούς μέσω Βουλγαρίας και μέσω ε, Αιγύπτου. Η χώρα σας όμως δεν βρίσκεται μόνη της, την στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, στηρίζουμε τη Βουλγαρία όπως και τα άλλα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής και τη βοηθάμε να διαχειριστεί, να ε, ελέγξει όχι μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά και τα σύνορα της Ευρώπης. Έχουμε παράσχει πολλή βοήθεια. Και θέλω να σας θυμίσω ότι όταν εγκαινιάσαμε την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, όλοι πήγαμε στο σημείο διέλευσης των σύνορων, ε, ε στα σύνορά σας με την Τουρκία, και ο νέος αυτός οργανισμός έχει ξεκινήσει τις εργασίες του και ξεκινήσαμε από τη Βουλγαρία. Στηρίζουμε τη χώρα σας και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε και στο μέλλον. Τελευταίο όμως και εξίσου σημαντικό, η Βουλγαρία έχει δεσμευτεί και η Βουλγαρία παρουσιάζει και αποτελέσματα. Η κυβέρνηση και οι αρχές έχουν πάρει στα σοβαρά, έχουν καταλάβει τη σημασία της αποστο... Ε, την αποστολή τους ως ε, υπερασπιστές των Ευρωπαϊκών Συνόρων. Ε, Μανώλης Κωστίδης από τον Sky. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή πολλές φορές έχω επισκεφτεί την Τουρκία. Ε, καταρχάς, είστε ικανοποιημένοι ε, με τη συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό, διότι ε, οι ροές έχουν μειωθεί από όσο βλέπουμε. Από την άλλη, πολλές φορές ε, που έχω επισκεφθεί και τους προσφυγικούς καταβλισμούς, οι Τούρκοι εκφράζουν ε, τις επιφυλάξεις για τη συμφωνία, διότι λένε τουλάχιστον ότι η Ευρώπη δεν τηρεί κάποια συμφωνηθέντα, όπως η Βίζα, όπως κάποια οικονομικά. Ε, ποια είναι η άποψή σας και πού θα οδηγηθεί αυτή η συμφωνία, αν υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες. Πρώτα απ' όλα, κύριε Κωστή, να σας πω ότι δεν πρόκειται για συμφωνία. Δεν είναι agreement σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Είναι statement διότι εάν επρόκειτο να συναυθεί μία συμφωνία θα έπρεπε αυτή να ακολουθήσει τη γνωστή διαδικασία εθνικά κοινοβούλια κλπ. Και νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ εκεί που φτάσαμε πριν από περίπου 17 μήνες. Τότε είχαμε περίπου 15.000 διελεύσεις μέσω του Αιγαίου προς την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδος. Το πόσο επιτυχής είναι η ευρωτουρκική αυτή δήλωση ως προς την εφαρμογή της αποδεικνύεται από τα νούμερα. Ο αριθμός αυτός τον τελευταίο χρόνο έχει πέσει κατά μέσον όρο στα 50 άτομα την ημέρα. Από την άλλη πλευρά οι ελληνικές αρχές οργανώθηκαν. Ναι, είναι αλήθεια ότι καθυστέρησε η Ελλάδα, αλλά με τη βοήθεια τη δική μας, την οικονομική, την πολιτική, σε τεχνογνωσία, σε experts. Σήμερα η Ελλάδα ελέγχει πλήρως τα ευρωπαϊκά, άρα και τα δικά της ε, σύνορα, με 100% ταυτοποίηση, δακτυλοσκόπηση και αναγνώριση όλων εκείνων που έρχονται στην Τουρκία. Τι προβλέπει όμως αυτή η ευρωτουρκική δήλωση. Προβλέπει ότι οι επιτροπές που έχουν συσταθεί από ελληνικής πλευράς στα νησιά, στα νησιά θα πρέπει να διεκπεραιώνουμε ακόμα με ταχύτερους ρυθμούς τα αιτήματα για την παροχή ασύλου που υποβάλλονται. Λέει λοιπόν η Τουρκία ότι εμείς είμαστε να πάρουμε πίσω όχι εκείνους που θα επιστρέψουν από την ενδοχώρα ή από την Ευρώπη, αλλά εκείνους που βρίσκονται στα νησιά. Σε κάποια στιγμή παρατηρήθηκε μια καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση είχε σαν αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός από ε, από μετανάστες ή πρόσφυγες, γιατί ακόμα δεν έχει ε, αποφασιστεί τι ακριβώς είναι, να είναι επάνω στα νησιά. Συνεπώς η ευρωτουρκική δήλωση λειτουργεί και λειτουργούσε μάλιστα πρέπει να πω ακόμα και κατά την διάρκεια του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία. Τι δείχνει αυτό την πραγματική βούληση της Τουρκίας να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Τα άλλα θέματα που θίξατε δεν αποτελούν μέρος, μέρος αυτής της δήλωσης. Το μόνο που έχει να κάνει με τη δήλωση είναι η οικονομική στήριξη με τα περίφημα 3 δισεκατομμύρια, τα οποία θέλω να διευκρινίσω για μια ακόμα φορά δεν δίνονται στην Τουρκία, αλλά μέσω των διεθνών οργανισμών και κυρίως του UNHCR, στο ειδικό φαντ που υπάρχει εκεί για να ε, διαχειρίζεται ε, θέματα όπως έχουν κάνει τη διατροφή, την ιατρική περίπτωση και άλλα των προσφύγων που ήδη βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος και που πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια. Συνεπώς, στο ερώτημά σας αν λειτουργεί αυτή η δήλωση, ναι λειτουργεί και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσει να λειτουργεί και στο μέλλον. Και εδώ ακριβώς είναι κατανοητό πόσο σημαντική είναι και η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και θέλω να πιστεύω ότι τίποτα δεν θα διασαλεύσει αυτήν την συνεργασία, γιατί είναι επόφελος, επαφελία, συγγνώμη, και της ε, Ευρώπης και της Τουρκίας και της Ελλάδας. Shall we take a last one or do you the last one? Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Εδώ. Παρακαλώ, Τάνια Μποζανίνο το Βήμα. Ε, η Γερμανία αποφάσισε να μειώσει δραστικά τους πρόσφυγες και μετανάστες που παίρνει κάθε μήνα από την Ελλάδα μέσω της οικογενειακής επανένωσης. Πώς το σχολιάζετε αυτό και πώς μπορούμε να πάμε προς τα εμπρός όταν πηγαίνουμε προς τα πίσω. εδώ και εδώ απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία επειδή καμιά φορά γίνονται και παρανοήσει. αξίζει να σα θυμίσω ότι μία από τι πρώτες χώρε που δημόσια δήλωσε ότι ανοίγει τι πόρτε τη για τι μετεγκαταστάσει από την Ελλάδα και από την Ιταλία, κυρίω όμω από την Ελλάδα, ήταν η Γερμανία. Με 500 περίπου άτομα ε, σε μηνιαία βάση. Αν αυτό που έκανε η Γερμανία το είχαν κάνει και οι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε λειτουργήσει με πληρότητα και αποτελεσματικότητα το ε, πρόγραμμα αυτό των μετεγκαταστάσεων. Δεν γινόμαστε στα πράγματα. Ακούσατε τι είπα προλίγου και στον συνάδελφό σας από την Ουγγαρία. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν το κάνουν. Συνεπώς αυτό λειτουργεί. Αλλά ως προς το συγκεκριμένο σημείο που θίξατε με την ερώτησή σας, επαναλαμβάνω ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η συνεργασία που ούτως ή άλλως είναι καλή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Το γεγονός ότι η Γερμανία θέλει να ε, ε, δέχεται και το έχει αποδείξει μέχρι τώρα είναι κάτι θετικό. Ε, και πρέπει να σας πω ότι είχα επαφή αυτές τις ημέρες και με τους δύο υπουργούς και με τον Γερμανό Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Ντεμεζιέρ και με τον Υπουργό Μετανάστευσης Ελλάδος, τον κυριο Μουζάλα οι οποίοι με διαβεβαίωσαν ότι αυτή η συνεργασία συνεχίζεται. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι έτσι πολύ απλά ε, να μην δημιουργούμε τέτοια θέματα και δεν αναφέρομαι στον τύπο, αναφέρομαι γενικώ στα όσα γράφονται κατά καιρού και ακούγονται. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και η Ευρώπη είναι εδώ, εγώ προσωπικά είμαι εδώ, οι υπηρεσίε μου, για να διευθετούν κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα που μπορεί να προκύπτει στην διαδικασία εφαρμογή αυτών των ε, προγραμμάτων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank very much your attention. Ε, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, σας εύχομαι καλή διαμονή στις εξωτικές Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε κύριε Επιτρόπη. Um, Το επίσημο κομμάτι του σεμιναρίου μας σήμερα λίγη εδώ. Θα σας δούμε στις 6 ώρα στο σαλονί των Ευρωβουλευτών κάτω. Ευχαριστώ.